Uh, I am very sorry to tell you that you should stop kissing. Ε, ζητώ συγγνώμη που θα σας ζητήσω να σταματήσετε τους χαιρετισμού και τα φιλιά, γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρία. μα. Ε, Καλώ ήρθατε λοιπόν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην συνεδρία τη Επιτροπής ΕΙΤΡΕ. Καλώς ορίζω και τι κυρίες και τους κυρίου φυσικά. Μπροστά μας και μπροστά σας Καταρχήν να, να, πω ότι ελπίζω να είχατε όλοι πολύ ευχάριστες ε, διακοπές ε, στις χώρες σας και να περάσουμε τώρα λοιπόν στην ημερήσια διάταξή μας όπου το πρώτο τη σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν σχόλια να θεωρήσω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε ως έχει. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Από εκεί και μετά έχουμε στο δεύτερο σημείο της ανακοίνωση του Προέδρου. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση, Ό,τι είχα να πω ήδη το είπα. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή κανόνες αστικού δικαίου για τη ρομποτική. Ε, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε θα τροφοδοτήσει την γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Γιούρη σε ό,τι αφορά την πρότασή της για τους κανόνες αστικού δικαίου για την ε, ρομποτική. Και η εν λόγω γνωμοδότηση θα εκφράσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτός ο ταχύως αναπτυσσόμενος τομέα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση στην στον παγκόσμιο τομέα της ρομποτικής. Ε, και βέβαια γνωρίζουμε ότι πολλά τμήματα αυτής της πολιτικής εδώ σχέση με τη ρομποτική ε, μπήκουν στις αρμοδιότητες της ΙΤΡΕ. Ε, ε, προφανώ οι κανόνε αστικού δικαίου αποτελούν αρμοδιότητα τη Επιτροπή Γιούρη, αλλά σχεδόν όλα τα υπόλοιπα που αφορούν αυτό το τομέα αποτελούν αρμοδιότητα τη Επιτροπή Ήτρε, όπω η βιομηχανική πολιτική, η χρήση των ρομπότ στο διάστημα, η ψηφιοποίηση και τα ζητήματα τηλεπικοινωνιών, όπω και η ε, πολιτική τη έρευνα και τη καινοτομία. Και αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση και την τηλεπικοινωνία. Ε, να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βέβαια σχετίζεται πολύ ε, με μια προηγούμενη γνωμοδότηση που είχαμε με την ε, συγκήτρια και αυτή τη γνωμοδότηση, κυρία Σκάλα. Οπότε να δώσω σε σένα το λόγο, Κάγια, ω την πρώτη λοιπόν ομιλήτρια μετά από το θερινό τη θερινή διακοπή εργασιών για το θέμα των κανόνων αστικού δικαίου σε σχέση με τη ροποδική. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε μου δίνετε για αυτή την τιμή αν θέλετε, αλλά αυτή την ε, πίεση εντό εισαγωγικών που μπαίνουν πρώτο λόγου Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το ζήτημα της ροποτικής και των σχετικών κανόνων αστικού ε, δικαίου, θεωρούμε ε, πως ε, η περαιτέρω ε, προώθηση αυτού του τομέα θα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητά μας και όχι η φόβη σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής γιατί έχουν γραφτεί πολλά σε σχέση με το μέλλον και το πώς αυτό θα διαμορφωθεί με βάση τα όσα θα λάβουν χώρα στη ρομποτική. Δεν έχουν αναφερθεί δηλαδή πολλά σε σχέση με τη συνεργασία που μπορεί να υπάρξει στο μέλλον ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ρομπότ. Και αυτό στο οποίο αναφέρομαι στη δική μου γνωμοδότηση εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλές μελέτες ότι θα μπορούσαν οι μικτές ομάδες ανθρώπων και ρομπόρ να είναι κατά 85% πιο παραγωγικές σε σύγκριση με ομάδες μόνο από ανθρώπους ή μόνο από ρομπόρ. Προφανώς ε, υπάρχουν εδώ και διαφορετικές μελέτες, αλλά ε, νομίζω πως ο στόχος είναι σαφής. Θα πρέπει να εστιάσουμε στη συνεργασία μόνο των ανθρώπων με τα ρομπόρ και όχι να εστιάσουμε στην αντικατάσταση των μεν από τους νέους. Ε, τώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δυνητικά εμπόδια που μπορούν να τεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της ρομποτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία μας, δηλαδή μέσω της, ε, ε, του εξυγχρονισμού της νομοθεσίας και μέσω της υιοθέτησης καταλήλων κατευθυντηρίων γραμμών για την πρόθεση εδώ της ανάπτυξης. Και προφανώ εκείνο που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ότι αν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή, δεν υπάρχει διασύνδεση, δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την ε, πρόθεση, γιατί η ρομποτική είναι δυνατή μόνο μέσω ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, real-time data flow. Ε, κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση και σε ό,τι αφορά τα δεδομένα ειδικότερα θα πρέπει να ζητούμε από την Επιτροπή να εξετάσει και τα ζητήματα διαλειτουργικότητας αλλά και τα, ε, τις ανοιχτές, ανοιχτού χαρακτήρα διαδικασίου. Οι, οι έξυπνες συσκευές και τα σχετικά δεδομένα θα λάβουν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία στο ε, μέλλον οπότε θα πρέπει να είμαστε ε, να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον τέτοιου είδους τεχνολογίες δεν θα είναι ε, περιορισμένες μόνο σε συστήματα, ε, σε υποσυγκεκριμένα περιορισμένα συστήματα ιδιοκτησίας. Ε, αυτά αναφέρω ε, εν και αναφέρω επίσης ότι ένα πιο ε, σε συστατικό ε, πλαίσιο κανονιστικό ουσιαστικά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ε, ε, προβλήματα για την πρόθεση. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει καινοτόμα συστήματα καταχώρηση των ευρεσιτεχνών του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στον κλάδο να αναλάβει ηγετικό τομέα σε ό,τι αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη η γνωμοδότηση αυτή που έχουμε ετοιμάσει το σχέδιο γνωμοδότηση εστιάζει στι αρμοδιότητε τη σύτρε σε σχέση με αυτό το ζήτημα, προκειμένου αυτέ να ληφθούν υπόψη στη γνωμοδότηση τη Επιτροπή ε, Γιούρη. Σα ευχαριστώ και αναμένω με ανυπομονησία την ε, συνεργασία μα. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο Κάγια, για αυτή την παρέμβαση και περνάμε τώρα στου εστιώδει συζητητέ μα εκ μέρου του ΕΛΚ Καλμπόνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε την Κάλια για αυτήν την εισαγωγική παρουσίαση και για τη συνεργασία μας, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία αυτή πριν από το καλοκαίρι. Ε, κάποια σχόλια θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι η περαιτέρω άπτυξη της αεροπολιτικής τεχνολογίας ε, σημαίνει και περισσότερες διαντιδράσεις, περισσότερες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Ε, δεύτερο σχόλιο. Ε, ζητήματα εκπαίδευσης, έρευνας ε, και ανάπτυξης και δράσης εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε σχέση με τη ρομποτική αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της σχετικής πολιτικής για τη ρομποτική. Τρίτο σχόλιο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής μέσω ε, συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και διεθνών επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα της ε, ρομποτικής. Ε, θα πρέπει να υπάρξει καινοτομία και να υπάρξει και μια ισχυρή κοινή αγορά και αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικούς στόχους ένα τέταρτο σχόλιο είναι ότι οι ε, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της, αυτού του νέου πλαίσιου, αν θέλετε, αυτή της νέας αγοράς, γιατί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ε, περαιτέρω προώθηση της ε, ε, και για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της αγορά, συγκεκριμένων υποτομέων τη αγορά. Οι ε, σχέσει ιδιωτικού δημοσίου τομέα, private public ε, partnerships μπορούν να συμπεριλάβουν τέτοιου είδου μικρομεσαίε επιχειρήσει και το Horizon 2020 ακριβώ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων στον χώρο τη ε, ρομποτική. Πέμπτο σχόλιο θεωρώ πω μέσω πρόθεσμα η ανάπτυξη του τομέα της ρομποτικής ε, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στους ε, ε, τομείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μεταπίση, όπως για παράδειγμα τομέα, τομέας, τομέας των υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Έκτος χώλιο, θεωρούμε πως η προώθηση της ρομποτικής θα πρέπει να συνδράμει και στην ανάπτυξη περισσότερο της χειρουργικής υψηλής ακρίβειας. Νομίζουμε πως με τέτοιες τεχνολογίες μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερο και θα πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη ε, υποστήριξη σε επίπεδο επιμελητία και στα ίδια τα νοσοκομεία. Και αυτό συμπεριλαμβάνει ε, το να λάβουμε υπόψη μα το πρώτο θα ελέγχουμε και πώ θα διαχειριστούμε τι ροέ δεδομένων μεταξύ ρομπότ και μεταξύ των ιατρών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέρνερ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάλλας για αυτή την ε, πολύ σύντομη αλλά και πολύ χρήσιμη Υπάρχουν ε, ακόμα πολλές ασάφειες ως το πώς θα εξελιχθεί μελλοντικά ο τομέας της ρομποτικής και σε ποιο βαθμό θα μεταλλάξει τις ε, αγορές. Ε, δηλαδή η, η ίδια η ρομποτική μεταβάλλει τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων και κατά συνέπεια έχει να κάνει πάρα πολύ και συνδέεται πάρα πολύ με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Ακριβώς δηλαδή κινείται στη, στον ίδιο άξονα με αυτή την ψηφιοποίηση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Ανάλογα λοιπόν με την μελέτη στην οποία βασιζόμαστε, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασία, αλλά και από την άλλη καταστροφή κάποιων θέσεων εργασία, μείωση του αριθμού των θέσεων εργασία. Και αυτή η τυχή δεν καλύπτει, κατά δική μου άποψη επαρκώ σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Επίση, το ζήτημα τη ασφάλεια θα πρέπει να καλυφθεί περισσότερο, γιατί κάθε τεχνολογικό άλμα, ειδικότερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, συνιστά και μεγάλη πρόκληση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων του και ε, των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ μπορούμε να παράσχουμε υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στι μικρομεσαίε Επιχειρήσει, επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που λείπει από, την, από αυτήν την γνωμοδότηση είναι η παγκόσμια πτυχή. Για παράδειγμα, η εξαγορά ε, της ε, κινέζικης, ε, του κινέζικου γίγαντα στην κούκα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί καταδεικνύει ότι η Κίνα έχει γνωρίσει την πάρα πολύ σημα... υψηλή σημασία, τη μεγάλη σημασία του τομέα της ρομποτικής οπότε ζητώ για μία ακόμα φορά από την Επιτροπή να αναπτύξει μία βιομηχανική πολιτική η οποία θα καλύπτει αυτούς τους πολύ σημαντικούς τομές για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε εδώ τις θέσεις εργασίας και τη διατήρησή του αλλά και τη διατήρηση του know-how της τεχνολογία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα εστιάσω λοιπόν ε, στι δικέ μου προτάσει ε, τροπολογιών σε αυτά τα ζητήματα που μόλι ανέφερα και χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε την κυρία Κάλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο ε, Σιλικιώτη εκ μέρου τη ΓΟΕ. Στον Πρόεδρε, ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Φοντιγιά για τη δουλειά που έκανε και την εισήγηση που κατάθεσε εδώ. Η τεχνολογική εξέλιξη, η ρομποτική και η αυτοματοποίηση υπόσχονται πολλά πλεονεκτήματα, Βράχει πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, για μας, για την ομάδα μας, είναι ξεκάθαρο πως για να έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα πρέπει η ρομποτική να αξιοποιηθεί με υπευθυνότητα για την εξυπηρέτηση των συμφρόντων και των αγκών της κοινωνίας, καθώς και για την ενίσχυση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό η αυτοματοποίηση και η ρομποτική να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Εξίσου σημαντικό είναι να ασφαλίσουμε πω ο τομέα τη ρομποτική θα στηρίξει το εργατικό δυναμικό, θα ενισχύσει τι ανθρώπινε δυνατότητε και θα δώσει νέα όθηση στη βιομηχανία. Ε, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυναμική που παρέχει η ρομποτική, ώστε να καλύψουμε κενά και αδυναμίε που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία. Η πραγματική οικονομία, θα έλεγα. Ιδιαίτερα στον νότο τη Ευρώπη, όπου α, σε αυτήν την περίοδο υπάρχει μια διαδικασία από βιομηχανοποίησης, είναι αναγκαίο να προωθήσουμε την καινοτομία στον τομέα της ρομποτικής, ώστε να στηριχθεί μια νέα εκβιομηχανοποίηση. Ε, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα ωφέλη της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης, πολλές φορές λόγω όχι επαρκό μέσο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσο θα έπρεπε ε, την ρομποτική. Ε, εάν όμω ε, τα κίνητρα είναι το αθόμητο κέρδο σε βάρο των ανθρώπων, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να καταπατηθούν ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίε και να προκληθούν σοβαρέ κοινωνικέ συνέπειε από τη χρήση τη ρομποτική. Γι' αυτό χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ε, απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ρομποτική θα είναι εργαλείο για την εξυπηρέτηση μονάχα των αναγκών του ανθρώπου και πρέπει να πω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και οι δικές μας οι τροποποίησεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. thank you much, Ευχαριστούμε πάρα πολύ συνάδελφε. Από την EFTD, ο κύριος Ταμπουράνο. Ε, Σας ευχαριστώ. Εμείς στηρίζουμε την γνωμοδότηση της συναδέλφου Κάλλας, αλλά θεωρούμε ότι σαν Ήτρε θα πρέπει ε, να ε, υπογραμμίσουμε, όπως έκανε και η Γιούρη, ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική υπηρεσία για την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ρομποτική, ρομποτική η οποία παίζει τεράστιο ρόλο στην ε, βιομηχανία. Και θα πρέπει οπωσδήποτε και η σχετική νομοθεσία να ευθυγραμμίσει ε, με τη, όπως άλλωστε το λέει και η κυρία ε, με τις ε, συγκεκριμένες ανάγκες και να σχετίζονται και να αναφέρονται οπωσδήποτε στην ψηφιοποίηση και την συνδεσιμότητα. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη ότι τα ρομπότ ενδεχομένως σχετίζονται και με σχέσεις με δημιουργία θέσεων εργασίας. Επομένως, θεωρούμε θεωρούμε ότι πέρα από ένα θέμα ε, αστικής ε, ευθύνης, ε, ασφάλειας δηλαδή, όπως ας πούμε για τα αυτοκίνητα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί και ένα είδος ταμείο πολιτών που θα στηρίξουν αυτούς τους εργαζόμενους που λόγω ακριβώς της διεύθυνσης χρήσης του ρομπότ θα χάσουν την εργασία τους. Νομίζω ότι αυτό το υπογράμμισε και η Επιτροπή Επιτροπή Γιούρη και εμείς αν θα πρέπει να το πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σα. Ε, η κυρία Κάπελ από την ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συμμερίζομαι την ε, άποψη της ε, κυρίας Κάλλας ότι το ε, σχέδιο γνωμοδότησης μας προς την ε, Γιούρη δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά περίπλοκο. Γιατί αν είναι πολύ περίπλοκο το μελλοντικό πλαίσιο ουσιαστικά θα έχει αναστατικό, θέλετε, αναστατική επίδραση στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ρομποτικής. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ όταν προτείνουμε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κατακνίξουμε ε, την καινοτομία, αλλά ούτε και τι δυνατότητε που δίνει το εταιρικό δίκαιο. Τώρα, εμείς τι βλέπουμε με επικριτικά στη γνωμοδότηση της ε, Γιούρη. Ε, τα ρομπότ να λάβουν ουσιαστικά μία ιδιότητα ε, προσώπου ε, νομικού δικαίου και να υπάρχει και ε, να έχουν νομική προσωπικότητα και να περιλαμβάνονται μέσα σε ένα μητρό τέτοιων ρομπότ. Είμαστε πολύ κριτικοί απέναντι σε αυτήν την πρόταση της Γιούρη, αλλά θα συμμετάσχουμε επικοδομητικά και θεωρούμε πως είναι σημαντικό το να υπάρξει μια τέτοια γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής Γιούρη, γιατί πραγματικά έχει ηγετικό ρόλο εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% της παγκόσμιας αγοράς ρομποτικής ε, συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει αυτό το μερίδιο να επεκταθεί ε, ακόμα περισσότερο μέσω μια επανεκβιομηχάνηση, αν θέλετε, όπω ήδη αναφέρθηκε από συναδέλφου. Ε, δηλαδή, ε, και αυτή η εξαγορά που έγινε του σχετικού ομίλου ήταν πάρα πολύ σημαντική και δεν ήταν τυχαίο ότι αναφερόταν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ε, στις, ε, στον τύπο και μια αντίστοιχη ε, ιαπωνική επιχείρηση ανέφερε ότι ε, θέλει να διπλασιάσει ε, τις δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,1 δισεκατομμύρια ε, ρομπότ έχουν εγκατασταθεί μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό ο αριθμό. Οπότε ε, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό ο ε, τομέα για, την, για τον βιομηχανικό κλάδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η συνεργασία στο μέλλον μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, ανθρώπων και ρομπότ, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να συμβάλλει και στην ε, βελτίωση των συνδικών εργασία, όπω έχουμε δει για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για παράδειγμα, έχουμε δει ότι μέχρι στιγμή η κατάσταση ανταλλακτικών ελαστικών σε πολυπαγκέ γινόταν μέχρι στιγμή από ανθρώπου, ενώ τώρα αυτή την εργασία την έχουν αναλάβει ρομπότ. Τέτοιου είδου παραδείγματα πώ να μα δείξουν πώ μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των συνδικών εργασία η ρομποτική στο μέλλον. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σάφχοζερ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω Ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω σε λεπτομέρειες ε, κατά την εξέταση αυτού του ζητήματος γιατί είμαι εισηγητής ε, για τις υπηρεσίες για τα cloud services και δεν μπόρεσα. Σε γενικές γραμμές οι αρχές μπορούν να είναι πολύ πιο χαλαρές γιατί ο προγραμματισμός θα γίνει στο πλαίσιο των cloud και συχνά στο λογισμικό χρήσης. Όσον αφορά τα ρομπότ, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ε, πολλαπλότητας ε, ε, καθηκόντων και αποστολών των ρομπότ. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και μιλάω κυρίως για τη βιομηχανία. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα εμπιστευτικότητας κρυπτογράφησης των δεδομένων γιατί διαφορετικά οι ξένοι ανταγωνιστές μπορεί να γνωρίζουν την τεχνολογική μας διαδικασία ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να διαφυλάξουμε αυτά τα δεδομένα σε σχέση με αυτό που ε, συχνά αποκαλούμε ανοιχτά δεδομένα. Η σημασία της Γερμανίας ε, ε, και της ε, προστιθέμενης αξίας ε, είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλη. Η Google και η Amazon επενδύουν πολλά, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια για το ζήτημα αυτό. Οι Κινέζοι επίσης το θεωρούν προτεραιότητα, αν δεν ε, είμαστε πρωτοστάτες στην τεχνογνωσία, ε, θα χάσουμε την ανταγνωστικότητά μας στο τέλο, στο, στο μακροπρόθεσμα. Αν χάσουμε αυτήν την τεχνογνωσία, θα ε, σημάνει καταστροφή κάτι τέτοιο για μας. γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Η Γαλλία βέβαια δεν είναι στο επίπεδο της ε, Γερμανίας ε, όσον αφορά το επίπεδο ε, είναι διπλάσια η ποιότητα της των γερμανικών ρομπότ και η Γαλλία δεν τα πάει πολύ άσχημα, που μας δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική είναι η δουλειά της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια τεχνογνωσία στην Ευρώπη εν, εν, εν, ενώπιον των ξένων ανταγωνιστών που δεν διστάζουν να καταστήσουν το θέμα αυτό άμεση προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. οποιαδήποτε όλες οι ερωτήσεις θα απαντηθούν γραπτώς ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν ε, ε, παρίστεται κανένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σήμερα εδώ. Γραπτός όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στις παρατηρήσεις και στις ερωτήσεις σας. Και το, για να φτάσουμε στο τέλος της συζήτηση αυτής, η εισηγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω Πολλοί από εσά είπατε ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εργασία και συμφωνώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τη ρομποτική. Όμω η Επιτροπή Απασχόληση ε, εκπονεί μια γνωμοδότηση επί του θέματο αυτού και όταν ε, το ε, συζητούμε το θέμα αυτό, έχω διαβάσει και πολλά σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα και είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα. Το ερώτημα είναι προς τα που κινούνται οι εργασιακές σχέσεις γενικότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, ε, σύμφωνα με μελέτες, 50% των ε, παιδιών ε, που γεννιούνται σήμερα δεν δουλεύουν στις, δεν θα δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν σήμερα, αλλά σε εντελώς νέες. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Η συνεργασία μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων θα δημιουργήσουν ενδεχομένως θέσεις απασχόληση που δεν γνωρίζουμε σήμερα. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην είναι το πιο συνετό Ούτως ή άλλως βέβαια η Επιτροπή Απασχόλησης απασχοληση ασχολειται λεπτομερέστερα με το θέμα αυτό και δεν είναι τη αρμοδιότητα τη δική μα επιτροπή ε, να ασχοληθούμε με τι εργασιακέ σχέσει. Εμεί επικεντρωνόμαστε περισσότερο στι βιομηχανικέ πτυχέ. Για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμφωνώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την εκμάθηση των μηχανών κλπ. Όσον αφορά ε, τώρα την υπηρεσία ε, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι η νέα υπηρεσία θα προσφέρει τίποτε το πολύ καλό. Ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη οργανισμοί που θα μπορούσαν να αναλάβουν ε, τη, τα ζητήματα που πρέπει να ε, καλύψουμε. Με χαρά θα περιμένω τη συνεργασία μαζί σας και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Ισηλήτρια. Να σας πω ότι 8 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, δηλαδή σε τρεις μέρες από τώρα. Μην καθυστερείτε. Ψήφο στην Ήτρε 10, ψηφοφορία στην Ήτρε, συγγνώμη, 10 Νοεμβρίου ε, και στην αρμόδια καθήλια επιτροπή Γιούρι 29 Νοεμβρίου, έτσι ώστε ε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ε, ψηφίσουμε ε, στις 10 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μπορέσει η Γιούρη να ψηφίσει στις 29 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως. Είμαστε άψογοι όσον αφορά το χρόνο μας. Ε, Προ μια περιφερειακή οικονομική σύγκληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα από πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο είχε η Ήτρε ε, προτείνει. Και τώρα πρέπει να δούμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για ένα από τα οχτώ προτινόμενα πιλωτικά προγράμματα σε σχέση με τον προηγούμενο προπολογισμό. Καλώς ορίσατε, καθίστε να σας πω δύο λόγια έτσι ώστε να σας υπενθυμίσω την κατάσταση και μετά ε, πρέπει να πω ότι θέλουμε να, έχουμε, να δούμε καλύτερα και από πιο κοντά ε, το συγκεκριμένο δοκιμαστικό σχέδιο Pilot Program TREC προς μια περιφερειακή οικονομική σύγκληση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το αναφέρουμε ως TREC εφ' ε, ξέρετε ότι ε, αυτού του είδους τα προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή καλή ευκαιρία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ήτρε γιατί καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα πιλωτικά προγράμματα, δηλαδή από την ώρα που ξεκινούν μέχρι την ε, δημιουργία του πραγματικού ε, προγράμματος και ε, μέχρι την χρηματοδότηση ενός grant στους grant holders οι οποίοι θα το αναπτύξουν. Ε, ποιο ε, είναι ο κύριος στόχος ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι ακριβώς ε, να φέρει σε επαφή τους πρωταγωνιστές και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών κλάστερ, καθώς επίσης και των τεχνολογικών κέντρων. Επίσης δε στόχο έχει την ανάπτυξη και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών κυρίως μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και μεταξύ λιγότερο αναπτυγμένων και προοδευμένων περιοχών. Η σύγκληση λοιπόν ε, προς ε, μια περιφερειακή ε, οικονομία. Αυτή η περιφερειακή οικονομική σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο στόχο. Ο κύριος στόχος, το δοκιμαστικό σχέδιο, το pilot project, το διαχειρίζονται δύο εταιρείες, τις οποίες θα θέλαμε ιδιαίτερως να έχουμε μαζί μας έτσι ώστε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο, πρώτα στον κύριο Χουάν Γουάς Κορομίνας, εκ μέρους του Grand Holder Eurecat, Τεχνολογικό Κέντρο της Καταλωνίας, δηλαδή από την Ισπανία, ο κύριος ε, Γουάσο Κοραμίνας είναι ε, Senior Public Program Area Manager στα αυτή τη Eurocat της Βαρκελόνης ε, της Ισπανίας. Η Eurocat είναι μια εταιρεία η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις αλλά και consulting όσον αφορά την ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας. Η πολυεθνική καθώς επίσης και πολυτομεακή ομάδα έρευνα ερευνητών ε, δουλεύει ε, σε πάνω από 160 ε, σχέδια και προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης. Είναι πάρα πολλά αυτά τα projects. Θα δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Κορομίνας. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, που μας δίνετε τον ε, λόγο, την ε, δυνατότητα δηλαδή να εκφραστούμε σαν ε, ε, κύριοι εκπρόσωποι αυτού του pilot project. Uh, uh, θα σας πω δύο λόγια όσον αφορά το πολιτικό μας πρόγραμμα και μετά ο κύριος Γκοτσάλντ από το άλλο πρόγραμμα θα πάρει το λόγο. Λοιπόν, εμείς ανταποκριθήκαμε ε, στην, ε, ε, στην πρόσκληση ενδιαφέροντος εκ μέρους της Eurocat, Eurocat η οποία έχει την έδρα της στην Ισπανία και η οποία ασχολείται με προχωρημένο manufacturing, κυρίως όσον αφορά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς ε, να δημιουργήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές τέτοιες ε, πρακτικές στην Ευρώπη. Τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή μπορεί κανείς να εξυγχρονίσει την, ε, τις παραδοσιακές μεταποιητικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Εμείς βασιστήκαμε σε δύο πυλώνες. Ε, ένας που μας επιτρέπει την χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σαν προσέγγιση για την προς την οικονομική ανάπτυξη κυρίως στις περιφέρειες της Ευρώπης και το ε, δεύτερο είναι μια ε, προσέγγιση ιδιαίτερης και εφιούς περιφερειακής εξειδικεύσεως. Εμείς συνεργαστήκαμε με την Καταλωνία, τον Βαρδίο, το Πάντε Καλέ και το α την ε, Νότια Ολλανδία. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, πρέπει να σας πω ότι προσπαθήσαμε να ε, καθορίσουμε ε, μια, ένα κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ των περιφερειών, ένα διαπεριφερειακό λοιπόν κοινό σχέδιο δράσης και ένα με αυτό σχετιζόμενο πρόγραμμα επενδύσεων. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσει κανείς τις εταιρικές σχέσεις, δηλαδή ποια θα είναι τα κλάστερς, ποια θα είναι τα τεχνολογικά ιστιτούτα, ε, τα οποία πρέπει κανείς να, ε, με τα οποία πρέπει να συνεργαστεί. Δηλαδή αυτά τα, αυτά τα ε, κέντρα τα οποία προσπαθούν να παράγουν χρήμα βάσει της υφιστάμενης γνώσης. Και βεβαίως, κατά δεύτερο λόγο, να δούμε ποιες είναι οι περιφέρειες με τις οποίες μπορεί να γίνει συνεργασία. Αυτό που έχουμε τώρα είναι αυτός ο κατάλογος που σας δείχνω με τα παραδοτέα ε, όσον αφορά κυρίως ανάπτυξη ε, υποδομών ε, δια σύνδεσης ε, ένα δεύτερο ε, στοιχείο είναι η ανάπτυξη ενός service model για την υποστήριξη της καινοτομία, Δεύτερον, ένα service mapping system, το οποίο θα είναι κοινό για όλες τις περιφέρειες, έτσι ώστε όλοι να δουλεύουν με το ίδιο μοντέλο, με το ίδιο εργαλείο, έτσι ώστε να υπάρχει και συγκρισιμότητα αφενός, αλλά και δυνατότητα μοιράσματος τεχνολογίας αφετέρου. Ε, φυσικά, ανάπτυξη νέων μοντέλων χρηματοδότησης. Γνωρίζουμε ποια είναι η δυσχέρεια όσον αφορά την χρηματοδότηση, κυρίως για το μεταποιητικό ιδιωτικό τομέα. Επομένω, πρέπει εδώ να υπάρξει ιδιαίτερη προσπάθεια και, τέ, και τέλος βεβαίως ένα ειδικό ε, σχέδιο, εξειδικευμένο σχέδιο επικοινωνίας. Ε, το πρόγραμμα θα τελειώσει ε, στο τέλος του τρέχοντος έτους. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διαπιστώσουμε βεβαίως ότι υπάρχουν διαφορετικές τυπολογίες clusters, ενώ στα τεχνολογικά κέντρα δεν παρουσιάζονται τόσο μεγάλες διαφορές. Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ των τεχνολογικών κέντρων, των clusters και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν ε, συγκεκριμένα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα κινητροδοτήσουν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα clusters, να δουλέψουν με τεχνολογικά κέντρα από διάφορα διάφορες ε, ε, περιφέρειες έτσι ώστε να ε, προσεγγίσουν με μεγαλύτερη εξειδίκευση τη στρατηγική στις διάφορες περιοχές. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η εμπλοκή των stakeholders, όπως ας πούμε είναι οι υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, ή ενώσεις βιομηχάνων λοιπά μπορούν να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και στην υπηρεσία των παρεχομένων περιεχομένων υπηρεσιών προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι τα τεχνολογικά κέντρα τείνουν να προσφέρουν παρόμοιε υπηρεσίε σε όλων των ειδών τη επιχειρήση, σε μικρέ μεσαίε ή μικρέ, ιδιαίτερα μικρέ, και ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό θα πρέπει ε, να το λύσουμε στο, ε, ε, στο μέλλον. Και τέλο, ότι οι μηχανισμοί περιφερειακής χρηματοδότησης τα στήριξη τη καινοτομία στι μικρομεσαίες αυτή τη στιγμή δεν ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το θέμα αυτό. Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να σας δείξουμε τώρα. Ε, βεβαίως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το πολιτικό μας πρόγραμμα και επομένως και η δράση μας. Αυτά ήθελα να σας πω για την ώρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ λίγο Πρόεδρο. Μας ε, ε, ευχαριστώ ευχαριστούμε ε, που μας τα είπατε αυτά και μας τα δείξατε κιόλας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντάνιελ Γκότσαλντ από την Insight Bavaria. Ο κύριος Κόρσταντ είναι Managing Director ε, της Insight Bavaria Σμέδρα στην Βαβαρία, στο Όμπενμπουργκ, της, στη Βαβαρία της Γερμανίας. Ε, είναι μια υπηρεσία που παρέχει υπηρεσίες και σχεδιασμό ε, και διαχείριση σχεδίων. Το Insight Bavaria είναι μια πρωτοβουλία του Cluster Chemi Bayern, CCB, ένα δίκτυο δηλαδή εταιριών και ε, ερευνητικών Ινστιτούτων ε, που σχετίζονται με την ε, χημική βιομηχανία της Βαβαρίας. Ασχολείται και με την χημική βιομηχανία αλλά επίσης και με άλλους βιομηχανικούς τομείς και ε, κάνει συνεργασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, σε ε, στο δικό μας ε, project εμείς ε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την εξή πρόκληση. Έχουμε τρεις διαφορετικές περιοχές. Έχουμε στις κάτω χώρες, μια συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε τη Βαβαρία και έχουμε και το Νότιο Τυρόλο. Οπότε προσπαθούμε να σκεφτούμε, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε μια κοινή πολιτική ε, για ε, νέα υλικά. Γιατί αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε για αυτέ τι τρει περιοχέ, ε, μπορούμε να το καταφέρουμε και σε σχέση με άλλε περιοχέ και με άλλα project. Αφού προσπαθούμε ακριβώ να αισθημάσουμε στην παγκοσμιοποιημένη ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια κοινά project ανάπτυξη. Βρέθηκα πριν από δύο εβδομάδε στην Φιλανδία. Και ενώ ε, δεν περίμενα εκεί ακριβώ να υπάρξουν τέτοιου είδου mega projects ε, πάντοτε με την ε, ε, εμπλοκή τη Κίνα. Μόλι έφτασα τελικά στη Φιλανδία για να δω το τι συμβαίνει εκεί, μου είπαν ότι είμαστε πολύ απασχολημένοι γιατί περιμένουμε και την κινητική αντιπροσωπή για να μα παρουσιάσει το project τη. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε λίγο στο περιφερειακό επίπεδο, να δούμε ποιε είναι οι έξυπνε στρατηγικέ εκπαιδεύσει διαφορετικών περιοχών, να ενώσουμε αυτέ τι περιοχέ μαζί και να δούμε τι μπορούμε να, να λάβουμε ω προστιθέμενη αξία από αυτό. Ε, και εδώ βέβαια πάντοτε προσπαθούμε να, έχουμε, να εστιάζουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά τα fine chemicals ε, μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε μια κοινή αλυσίδα παραγωγής, δηλαδή το κάμελο να ξεκινάει αυτή την παραγωγή μετά στην Βαυαρία να γίνεται υπεραιτέρω επεξεργασία και μετά να εφαρμόζεται για παράδειγμα στο νότιο Τυρόλο η χρήση τέτοιων, τέτοιων χημικών σε συγκεκριμένε περιβαλλοντικέ συνθήκε. Ε, για παράδειγμα, στον ε, τομέα των καθαρών τεχνολογιών, ε, έχουμε δηλαδή σε διαφορετικέ αλυσίδε παραγωγή προστιθέμενη αξία αυτή τη δυνατότητα και αυτόν τον στόχο τον εξετάσουμε τελικά. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια συνεργασία. Έχουμε αξιολόγηση ε, τη όλη διαδικασία. Έχουμε κοινέ αγορέ, κοινή δραστηριοποίηση. Αν υπάρχουν αυτέ τα προαπαιτούμενα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλάστερ. Ε, εάν δεν υπάρχουν αυτά τα προαπαιτούμενα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω να το ξεχάσουμε. Αν λείπει όμως ένα από τα προαπαιτούμενα, τότε έχουμε τις ε, στρατηγικές επενδύσεις ε, κλειδιά όπως λέγονται, key strategic investments, ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα βιοηλικά ε, που χρησιμοποιούνται ε, στον ιατρικό τομέα, για παράδειγμα για κάποια εμφυτεύματα ή για παράδειγμα χρήση τρισδιάθατων εκτυπωτών για τέτοιου είδους εμφυτεύματα. Εάν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τέτοια ε, εκτύπωση τέτοιων ε, τρισδιάστατων ε, προϊόντων όπως αυτά προβλέπονται από μια άλλη περιοχή στο Νότιο Τυρόλο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι επιτυχημένο κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε κάποιες στρατηγικές επενδύσεις κλειδιά για να μπορούμε να επιτύχουμε όλα τα προαπαιτούμενα που επιτρέπουν αυτήν την συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Και λέμε ότι θέλουμε οι επενδύσεις αυτές να εστιάζονται ακριβώς στα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν την παραγωγή αξίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Για παράδειγμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, ε, ε, και αυτό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο επενδυτέ, είτε είναι από τι ΗΠΑ, Πολιτείε, είτε από, από την Κίνα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε ω βασική επένδυση για να ε, θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την ε, διαπεριφερειακή αν θέλετε παραγωγή αξίας. Ε, όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα ούτω ή και στο διαδίκτυο για να δούμε το τι μπορούμε να, να πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο και αλλού. Για παράδειγμα να πάρουμε μία, ένα μηχάνημα ε, ένα μηχανισμό αν θέλετε, ο οποίος, μια φόρμουλα η οποία θα παίρνει μια ιδέα μια παραγωγή σε μια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωση και θα μετατρέπει σε μια επένδυση, σε μια πρωτοβουλία, σε μια άλλη περιοχή. Και αυτό νομίζω μπορεί να μας επιτρέψει ε, να έχουμε μια τέτοια συνεργασία και εμείς αυτόν τον μηχανισμό τον ε, ονομάζουμε ω επιταχυντή διευρωπαϊκών επενδύσεων. Αυτό που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει είναι να πάρουμε αυτό το μηχανισμό και να τον συνδυάσουμε με ε, ε, χρηματοδοτήσεις, με επενδύσεις ε, δηλαδή. Γιατί μέχρι στιγμής τέτοιου είδους μοντέλα έχουν συμμοσιμοποιηθεί σε πολύ σε διαφορετική ποιότητα, αν θέλετε, χαμηλότερε σε ποιότητε επενδύσει, για παράδειγμα, και ένα νέο καζίνο ή κάτι τέτοιο. Εάν δούμε ε, πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιου είδου επενδύσει διαπεριφερειακέ σε πραγματικά παραγωγικά project, μπορούμε να δούμε το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Ε, για παράδειγμα, υπάρχει μια τέτοια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τι ε, διαπεριφερειακέ συνεργασίε. Και με τέτοιου είδου επενδύσει μπορούμε και εμεί να επιτύχουμε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε πω ε, ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορέσει να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τη δική σα ε, εδώ Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά τηρήσατε το χρόνο σας με τρομερή ακρίβεια. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μαραγκάλ, ο οποίος ε, ήταν ένας από τους εμπνευστές ε, της ιδέας αυτής, του πιλωτικού ε, προγράμματος στην Επιτροπή μας και εξ όσων γνωρίζω θα θέλατε να μας δείξετε και διαφάνειες. Μπορείτε, μπορείτε. Έχετε το λόγο κύριε Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα κατανοήσετε αυτό, αυτή την ε, γραφική ε, παράσταση Μπορείτε βεβαίω να τη χρησιμοποιήσετε και να τη δείξετε σε όποιον ε, ενδιαφέρεται. Είναι η σχέση μεταξύ της ε, παραγωγικότητας ε, και του κόστους εργασίας αναώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015. Απλώ και μόνο για να δει κανεί τη σχέση μεταξύ αυτών ε, των δύο ε, τιμών. Ε, τα πράγματα έχουν όπως φαίνεται στην γραφική αυτή παράσταση. Θα ήθελα να συνεχίσω στα ισπανικά τώρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, τον κύριο Σκατίνα και την Dizzy Growth Να τους ευχαριστήσω και κυρίως να ευχαριστήσω βέβαια τους δύο πρωταγωνιστές της ημέρας που ήρθαν εδώ ως εκπρόσωποι της Insight ε, Bavaria καθώς επίσης και τον Juan Guas από την ε, Καταλωνία. Η Βαβαρία και η Καταλωνία λοιπόν. Αυτές οι δύο περιοχές δεν είναι τυχαίο που έχουν δημιουργήσει τέτοια κλάστερς ε, γιατί οι τεχνολογικές ε, εξελίξεις αυτών των ομόσπονδων κρατηδίων και των αυτονόμων περιοχών είναι κάτι επιβεβαιωμένο πλέον. Δεν θα μιλήσω πολύ αλλά να πω κύριε Πρόεδρε ότι η επιτυχία του πολυπλωτικού προγράμματος που μέσω αυτών των δύο εμπειριών παρουσιάζεται σήμερα καταδεικνύει ότι είμαστε ε, σε θέση εμείς σαν Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σαν ε, Επιτροπή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε ικανοί λέω να βοηθήσουμε περιοχές οι οποίες είναι περισσότερο αναπτυγμένες σε τον ένα ή τον άλλο τομέα να τις διασυνδέσουμε με άλλες περιοχές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα μέσω της αύξησης της ε, παραγωγικότητας μέσω της αποδοχής αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης να βελτιώσουν την ε, απόδοσή τους γιατί εδώ το ζητούμενο δεν είναι η μείωση ε, του μισθολογικού κόστους μονάχα αλλά να έρχονται σε επαφή οι περιφέρειες μεταξύ τους έτσι ώστε η μία να μαθαίνει από την άλλη έτσι ώστε η μία να επηρεάζεται στις επιλογές της από την άλλη έτσι ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και βεβαίως εγώ είμαι πεπισμένος ότι όταν μιλάμε για, ε, ε, ε, για βιομηχανική πολιτική, αυτό το μεγάλο απόντα δηλαδή τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτό το ευρωπαϊκό παράδοξο, δηλαδή εξαιρετικό επίπεδο έρευνας αλλά πολύ χαμηλότερο επίπεδο δυνατότητα δυνατότητας μετατροπής αυτής της έρευνας υψηλού επίπεδου σε εξίσου υψηλού επίπεδου καινοτομία, αυτό το ε, παράδοξο ελπίζουμε ότι με τέτοιου είδους προγράμματα θα ε, λυθεί. Είναι σημαντικό και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Οι χώρες που δεν αναφέρονται Δέκα χώρες ε, μέλη δεν αναφέρονται στην ε, ε, γραφική αυτή παράσταση. Έχετε απάντηση γι' αυτό. Νομίζω όλες αναφέρονται 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από την Eurostat τα στατιστικά στοιχεία. Είναι επίσημα τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για αυτή τη γραφική παράσταση. Λογικά πρέπει να αναφέρονται όλα τα κράτη-μέλη περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως να αναφέρονται τα κράτη-μέλη, αλλά όχι η σχέση κάθε φορά. Σε αυτό μπορεί να έχετε δίκιο. I've got here, Okay. Ίσως είναι διαφορετικό αυτό που, έχετε, που μας δείχνετε στην οθόνη από αυτό που έχω μπροστά μου. Ο κύριος Μαραγκάλ. Ναι, βεβαίω, να σα δώσω όλα τα στοιχεία, τον πλήρη φάκελο, αν θέλετε. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο, ρωτάει πρόεδρο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τοκάρσκι, ε, που είναι ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Grow, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να σχολιάσουμε αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαστε πολύ ευγνώμονε στην Επιτροπή σας για την υποστήριξη από την πρώτη μέρα για την υλοποίηση αυτών των projects και ειδικότερα ε, προς τον κύριο Μαραγκάλ για την δική του συνεισφορά. Αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια ευρύτερη προοπτική. Θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα δύο προγράμματα για την ε, αναβάθμιση της προσέγγισης τύπου κλάστερ, ε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε μια νέα δραστηριότητα που θα αρχίσει το 2017 υπό το κόσμο για να διαμορφωθεί και να ε, αναβαθμιστεί μια ένα πρόγραμμα για την έξυπνη επένδυση, της μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, δημιουργήσαμε λοιπόν ε, αυτήν τη νέα ε, δια, δραστηριότητα η οποία θα αντιγράψει ουσιαστικά αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα με πολλούς τρόπους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ήδη, η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί ε, θα συμπεριληφθούν πολύ σημαντικά τεχνολογικά Ινστιτούτα που θα υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ώστε να μπορούν διαρθρωτικά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό το ε, προϋπολογισμό του κόσμου 2 εκατομμύρια για το 2017 και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν 5 κλάστερς για διάφορα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν κλάστερς από τουλάχιστον μία περιφέρεια ε, ή μία περιφέρεια σε μετάβαση. Θέλουμε να υπάρχει μία διαδικασία αμοιβαία εκμάθηση στο πλαίσιο τη προσεγγιση αυτη Αυτό που επιση κάνουμε παράλληλα είναι προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τι περιφερειακέ αρχέ στην προσέγγισή μα. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μαζί με την Γενική Διεύθυνση Regium μία πλατφόρμα για αυτήν την FEE e επένδυση ε, οι περιφερειακές αρχές θα μπορούν ε, να προσφεύγουν στην πλατφόρμα για ε, κατά παραγγελία καθοδήγηση και συμβουλές και αυτό θα βοηθήσει την ευρύτερη εταιρική σχέση γενικότερα. Ε, εξετάσαμε αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα για να δούμε αν υπάρχουν κάποια διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Για παράδειγμα, συζητούμε με τους εταίρους ε, στα προγράμματα πώς ε, μπορούν τρίτα κλάστερ σε σχέση με τη μεθοδολογία ή με τη συνεργασία, πώς μπορούμε δηλαδή να βελτιώσουμε ε, ε, την κατάσταση, ε, εργαστήρια ή τεχνολογικά Ινστιτούτα, εγκαταστάσεις, μηχανισμοί να είναι διαθέσιμα και σε άλλα κλάστερς. Υπάρχουν δηλαδή πολλές δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε, να συνοψίσετε τη συζήτηση. Κάποιες συμπερασματικές λοιπόν παρατηρήσεις. Ε, ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση, γιατί μιλήσατε και για άλλες περιφέρειες και για το όφελος ε, για άλλους εταίρους. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να είναι διαθέσιμο για κάθε, να είναι διαθέσιμο για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν αυτά είναι προγράμματα στα οποία ε, μεγιστοποιούν το δυναμικό μία και μόνο περιφέρειας, δεν θα λειτουργήσει. Θέλουμε να είναι διαθέσιμο για όλους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση και θα είναι έτσι πολύ πιο δυνατό το εργαλείο αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε ιδιαίτερω από τις αρχές του επόμενου έτους. Ε, σα ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ ιδιαίτερω την Επιτροπή σα γιατί κατέστησε δυνατή ε, αυτή την προσπάθεια. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα, για τα προγράμματά σα, για την ε, παρουσίαση που κάνετε και για τα καλά αποτελέσματα που μα έχετε παρουσιάσει. Uh, Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε, δεν έχουμε πολύ κόσμο εδώ, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, δυστυχώς λέει ο Πρόεδρος. Θα ξεκινήσουμε, άσε που έχουμε καθυστερήσει κιόλα. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ερώτηση Είστε ευτυχεί που ξαναγυρίζετε στο κοινοβούλιο. Απαντήστε λοιπόν ψηφίζοντας ναι, όχι. Άρχεται η ψηφοφορία από αυτού του σημαντικού ερωτήματος. Ψήφισαν όλοι. Closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, φαίνεται ότι οι περισσότεροι είναι πανευτυχεί. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο το αποτέλεσμα. Πέραν πάση προσδοκίας. Λοιπόν, αρχίσουμε τώρα. Έχουμε έναν κατάλογο ψηφοφορίας. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Νίκολας Μπέι. Ευθύνη. Αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τροπολογία 20, ονομαστική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ η τροπολογία 20 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 25. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά αποχές καλύτερα να επαληθεύσουμε. Ελέγχουμε λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία την τροπολογία 21. Πέρας της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 22, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια ψηφοφορία, δεκτή η τροπολογία. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 23. Πέρα στις πληροφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές. Καλύτερα να το ε, επαληθεύσουμε. Επαλήθευση λοιπόν διελεκτρονικής πληροφορίας τροπολογία 26. Πέρας της πληροφορίας και η 26 27 διονομαστικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά. Καλύτερα να επαληθεύσουμε. 31. Ηλεκτρονική ψηφοφορία από τις τροπολογίες 31, πέρας της ψηφοφορίας, απερίφθη. Τροπολογία 32, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 διονομαστικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και γίνεται δεκτή η τροπολογία 35. 36 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την τροπολογία 36. πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές. δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 37. Πέρας της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ε, ελέγξουμε καλύτερα, δεν θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 39 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορία και γίνεται δεκτή η τροπολογία 39. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 40, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 42 υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον δεκτή, ναι. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 45 καταπίπτει, διότι η 37 είχε εγκριθεί, τροπολογία 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51, 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 52 άρχεται. Πέρας. Γίνεται δεκτή η τροπολογία 52. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 56, 55 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα. Συμβιβαστική 1, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απερίφθη. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 4 υπέρ κατά Καλύτερα να επαληθεύσουμε, ε, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 4, πέρας της ψηφοφορίας και και απερίφθη. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 12, κατά, Καλύτερα να ε, ε, ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 12. Τροπολογία 12. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 διονομαστικής κλίσεως άρχεται Πέρα της ψηφοφορίας και απερίφθη. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται τελική ε, ε, ψηφοφορία διηλεκτρονικής ε, ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε για την τελική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Επομένως δεν, έχουμε, δεν θα έχουμε ε, δι, της δικής μας Επιτροπής ε, ε γνωμοδότηση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διακυβερνητικέ συμφωνίε και μη Συγγνώμη, όσον αφορά την ευθύνη, την αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τι ευράκτητε δραστηριότητε εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν θα υπάρχει γνωμοδότηση τη ΙΤΡΕ. Έληξε λοιπόν η ψηφοφορία και περνάμε εις το σημείο 6. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε ιδιαίτερους ήσυχοι και σιωπηλοί κατά την έξοδό σας, εάν θέλετε βεβαίως να εγκαταλείψετε αυτή την αίθουσα. Ισχύει για όλους σας αυτό. Mr. as well. Christianis. Κύριε Κάριντς, αυτό ισχύει και για σας που λέω. Okay, so let us start. Let us start then. Εντάξει, να συνεχίσουμε λοιπόν. Είμαστε στο σημείο 6 τη Μεσαία Διατάξεω. Θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διακυβερνητικέ συμφωνίε και μη δεσμευτικά μέσα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και κατάργηση της απόφασης 94. Ε, να σας πω ότι αυτή η πρόταση κανονισμού ε, αποτελεί μέρος της δέσμης ε, για την ασφάλεια της ενέργειας που σκοπό έχει να δημιουργήσει ε, μια πιο δυναμωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας και να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και αυτό βεβαίως ε, θέλει να διασφαλίσει και την συμμόρφωση των ε, διακυβερνητικών συμφωνιών με, τον, ε, με την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς επίσης και να ενισχύσει τη διαφάνεια των συμφωνιών, καθώς επίσης και να αυξήσει την σχέση κόστους απόδοσης της παροχής ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμείς ε, πρέπει να πω ότι ο εισηγητής μας μας είχε παρουσιάσει την έκθεσή του τον Ιούνιο και είχε προτείνει 27 τροπολογίες, αλλά έχουν προσθεθεί και άλλες 203 τροπολογίες. Στόχος της σημερινής συζήτησής μας λοιπόν είναι να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες ε, πριν από την ε, διαδικασία εξέβρεσης ε, συμβιβαστικών λύσεων και τροπολογιών. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση δίνοντας πρώτα το λόγο στον εισηγητή, μετά στους σκιώδεις εισηγητές, έτσι να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε προς συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο συνάδελφος Τζισλούαφ Κρασνοντέψκι από την ECR είναι εισηγητής μας. Και σας δίνω το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, 203 ε, τροπολογίες ε, κατατέθηκαν. Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά όχι Έχουμε δει και χειρότερα. Προγραμματίζουμε μία ε, συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ενδεχομένως να είναι διαφορετική η ημερομηνία από αυτή που σας έχει γνωστοποιηθεί. Σήμερα ε, στείλαμε τις ε, προτάσεις συμβιβαστικών τροπολογιών και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι Κανονικά έπρεπε να ψηφίσουμε 13 Οκτωβρίου για την έκθεση αυτή. Όσον αφορά στις τροπολογίες, ε, θα μπορούσα να πω ότι το περιεχόμενο κινείται προς την αύξηση των δικαιωμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελέγχει τις ε, διεθνείς συμφωνίες υπάρχουν ε, συνάδελφοι που είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι από μένα και νόμιζα ότι ήμουν αρκετά φιλόδοξος στο πλαίσιο των τροπολογιών αυτών λοιπόν αν εγκριθούν η έκθεση πηγαίνει πέρα από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι, υπάρχει μία εντύπωση ότι ε, τα δεσμευτικά μέσα ε, ως τώρα δεν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι ε, που πρόσκυνται στην αριστερά και στη δεξιά και έχουν πολύ αποκλίνουσες απόψεις. Νομίζω πάντως ότι υπάρχει μία πλειοψηφία σε σχέση με την ε, απαλλαγή των διεθνών ε, ε, συμβάσεων και όχι τόσο των κρατικών συμφωνιών, των συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών. Το ζήτημα Αφορά και τα μη δεσμευτικά μέσα, ωστόσο. Οι συνάδελφοι σε γενικές γραμμές θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιορισμός ή ένας έλεγχος εγγράφων που δεν συνιστούν συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι από νομικής απόψεως το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των διεθνών συμφωνιών. Υπήρχε και μία πρόταση ελέγχου των συμφωνιών αυτών, στις οποίες τα μέρη, ε, τα συμβαλόμενα είναι όχι μόνο κράτη-μέλη, αλλά και επιχειρήσεις ε, που ελέγχονται κυρίως ε, από ε, τα κράτη. Σύμφωνα λοιπόν ε, και με την άποψη του Συμβουλίου, εμείς διαφωνούμε με ε, το να αφορά αυτό μόνο ε, δεσμευτικά μέσα. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος όχι μόνο βάση του ενωσιακού δικαίου, αλλά και βάση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Ένωσης και της Ενεργειακής Στρατηγικής. Θα μπορούσα να πω με αρκετή αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό αποτελεσματικό και ταχύτατο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης ε, των τροπολογιών. Από ό,τι κατάλαβα έχετε ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Τώρα να περάσουμε στους σκιώδεις εισηγητές εκ του ΕΛΚ, ο κύριος Ρούτσεφ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι, εγώ συμφωνώ με την πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση που ακολουθεί ο κύριος Κρασνοδέμσκι για την νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, για τη συνεισφορά τους, πάνω από 200 τροπολογίες. Έχοντας διαβάσει όλες αυτές τις τροπολογίες, θα ήθελα να τονίσω αρκετά ε, ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν πολύ λεπτομερώς στη μελλοντική εργασία μας. Καταρχάς, ε, κάποιες κόκκινες γραμμές πρέπει να γίνουν σεβαστές, ειδικότερα όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να αποφασίζουν τη δική τους ενεργειακή πολιτική πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία με τα, με τα κράτη-μέλη, με τις ε, ε, αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών. Πρέπει να γίνει σεβαστή η ε, επικουρικότητα και η αναλογικότητα και νομίζω ότι είναι προ συμφέρον των κρατών μελών ε, να, η εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τους ε, συνεπικουρεί και γι' αυτό νομίζω ότι ε, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερβαίνει τις κόκκινες γραμμές για τις οποίες μίλησα προηγουμένως και πρέπει να συμμετέχει μόνο κατόπιν εγκρίσεως των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Όσον αφορά τα μη δεσμευτικά μέσα τώρα, κατά την άποψή μου, τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να ε, υποβάλουν τα μη δεσμευτικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί νομικώς δεν είναι δεσμευτικά ακριβώς και συνεπώς τα μέσα αυτά δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από την απόφαση αυτή. Η υποβολή των μέσων αυτών θα έπρεπε να παραμένει εθελοντική, προαιρετική. Ε, διαφορετικά νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο διοικητικό άχθος και αυτό δεν είναι κάτι το έφικτο. Υπάρχουν φόβοι ότι τα κράτη-μέλη θα περάσουν από τις διακυβερνητικές συμφωνίες σε μη δεσμευτικά μέσα. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί υπερβολή. Σε κάθε περίπτωση, οι προθέσεις ε, των διαπραγματευτικών μερών θα καταλήξουν ε, σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, αν πρόκειται για πραγματικές διαπραγματεύσεις. Τρίτον, ας ε, είναι ε, τα πράγματα πιο σαφή με ε, πιο ακριβή ορισμό του τι είναι διακυβερνητική συμφωνία. Οι συμφωνίε για ενεργειακό ανεφοδιασμό και ενεργειακή υποδομή με δεσμευτικό χαρακτήρα μπορεί να επηρεάσουν το, την εσωτερική ενεργειακή αγορά ενός κράτους μέλους. Τέταρτον, κύριε Κρασνοντέμσκι, είπατε όσον αφορά τον περιορισμό της εκ των προτέρων κοινοποίησης ε, μόνο για ε, τις συμβάσεις που αφορούν τον το αέριο, τον τομέα του αερίου, νομίζω ότι αυτό αφορά το αέριο, γιατί στο πετρέλαιο έχουμε υποδομή που θα μπορούσε να επηρεάσει, να επηρεάσει την εσωτερική ενεργειακή αγορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μια διατύπωση να ε, πείσουμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει και εκείνο. Και τέλος, τα κράτη-μέλη πρέπει να κοινοποιούν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των προτέρων ε, τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, γιατί αυτό συνάδει απολύτω με τους στόχους της ε, Ενεργειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα ως προς την αύξηση της ενεργειακής, του ενεργειακού ανεφοδιασμού και επίσης συνάδει και με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μπαλτσίτης εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εξαιρετική είναι η δουλειά του. Είναι πολύ ε, δύσκολη ε, η θέση του όσον αφορά την υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει ένα αποτελεσματικό μέσο, αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών για τις ε, διακυβερνητικές συμφωνίες. Εγώ και ο δισηγητής θα ήθελα και εγώ να το τονίσω αυτό. Έχω εξετάσει όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες και μπορώ να πω ότι έχει καταφέρει ο εισηγητής να διατηρήσει τις βασικές προτάσεις που θα ενισχύσουν την ε, ε, ενεργειακή μας ε, αγορά. Όσον αφορά τα μη δεσμευτικά μέσα, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον, εκ των προτέρων, στην εκ των προτέρων, εκ των αξιολόγηση και συμφωνώ ότι με την ιδέα της πλήρους ενημέρωσης για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τώρα για τη, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαπραγματεύσεις Σωστή είναι αυτή η διάσταση και έχει ενισχυθεί στη συμβιβαστική τροπολογία 4 όπου θεωρείται υποχρεωτική η συμμετοχή αυτή, αν οι διαπραγματεύσεις καλύπτουν το 20% του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Επίσης, Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που οι διακυβερνητικές συμφωνίες στο μέλλον θα κρίνονται από το περιεχόμενό τους και όχι τόσο από τη μορφή τους. Αυτό αναφέρεται στην βαστική 1. Και θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Ελπίζω πραγματικά ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το περιεχόμενο ε, της έκθεσης αυτής είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας βοηθήσει στην ενίσχυση της ενεργειακής μας αγοράς στο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, ε, Mr. Palunder, replay... Ο κύριος Παλούντερ ε, αντικαθιστώσε τον κύριο Τάραντερ εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω πως ε, δεν μπορεί κανένας ε, να τονίσει επαρκώς ε, την σημασία των τέτοιων ειδικών συμφωνιών για την καλή, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι τα σημερινά συστήματα θα πρέπει να βελτιωθούν και εγώ συμφωνώ με αυτήν την διαπίστωση και θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων δεν παρακολουθεί απλώς τα πράγματα βοήθητη, αλλά ότι πραγματικά έχει τα εργαλεία στη διάθεσή της ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που χρειάζονται και οι πολίτες της. Ε, βλέπω με χαρά ότι υπάρχει ευρύτατη ε, υποστήριξη απέναντι σε αυτή την πρόταση, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα με η Επιτροπή να συμμετέχει στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών, αλλά θα πρέπει, should, να συμμετέχει σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, ώστε να μπορεί πράγματι να διασφαλίζει την ε, ασφάλεια του ενεργειακού ε, εφοδιασμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακρίνει ποιε είναι οι σημαντικές ε, συμφωνίες ε, και να επιλέγει να είναι παρούσα. Κατά τη δική μα άποψη πρόκειται για τις συμφωνίε εκείνε, οι οποίες ε, αφορούν το 20% των κάλυψη τη κάλυψη των αναγκών για τη συγκεκριμένη πηγή ενέργειας των 100 μελών που τη συναπτούν. προκειμένου να, να κλείσουμε εδώ παραθυράκια ε, στους νόμους, ε, δηλαδή ε, μέσω της, το να παρουσιάζεται μια διακυβερνητική συμφωνία με τη χρήση μιας εταιρείας η οποία όμως στην πραγματικότητα ε, κατέχεται ή βρίσκεται υπό τον ολεχο της, ε, του κράτους ε, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη δυνατότητα να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ έχουμε και το παράδειγμα για παράδειγμα της ρωσικής Κασπρόμα αφού αυτή έχει την δυνατότητα να συνάπτει τέτοιου είδους διακυβερνητικές συμφωνίες. Τώρα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τα όσα διαβάζουμε από τους συναδέλφους είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει πολύ επικοδομητική συζήτηση εδώ και ότι θα μπορέσουμε και να περάσουμε ένα πολύ εμφατικό θετικό μήνυμα από την πλευρά του ε, Γενοβουλίου και ε, αναμένουμε βέβαια την συνεργασία, επικοδομητική συνεργασία που θα έχουμε με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίρνινγκ που αντικαταστά η κυρία ε, Μίναρ εκ μέρους των φιλελεύθερων της Άντε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω σε και αισιόδη εισηγητέ ε, για την πάρα πολύ συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό το ε, φαντινό. Νομίζω πω ε, το σχέδιο τη έκθεση από την πλευρά του εισηγητή ήδη καλύπτει μία σειρά από σημαντικά στοιχεία προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλο που θα παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τη σύναψη τέτοιων διακυβερνητικών συμφωνιών. Εάν θέλουμε πράγματι να δημιουργήσουμε, να εδραιώσουμε μία ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια, θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι και οι διακυβερνητικέ συμφωνίες οι οποίε συνάπτονται συμμορφώνονται με το κανονιστικό πλαίσιο Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες, με τους μακροπρόθεσμους στόχους ε, στο πλαίσιο της σχετικής ε, πολιτικής ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει και κατάλληλη ανάληψη ευθύνης για την επίτευξη των σχετικών στόχων πολιτικής. Συμφωνούμε επί μία σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εξάντε εκ των προτέρων αξιολόγηση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, και επιβολή συμπληρωματικών ε, ρητρών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλλει πράγματι στην αύξηση τη διαφάνεια αλλά και στην αυξημένη συμμόρφωση με το δίκαιο τη Ένωση. Επίση, προτείνουμε μία σειρά από σημεία τα οποία θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το σχέδιο γνωμοδότηση και θα δώσουν ακόμα περισσότερε ε, δικαιοδοσίες εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο ακόμα στοιχεία τα οποία προτείνουμε είναι να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγηση όχι μόνο διακυβερνητικών συμφωνιών, αλλά και μη δεσμευτικών ε, μέσων μέσω εξάρτητη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε όμω παρόλα αυτά ότι κάθε αξιολόγηση από την πλευρά Επιτροπή δεν θα πρέπει να προδικάζει το ε, περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών. Το μόνο που θα πρέπει να κάνει αυτή η αξιολόγηση είναι να εξετάζει κατά πόσο η λόγω συμφωνία συνάδει ή όχι με το ε, δίκαιο τη Ένωση. Επίση, θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στι διαπραγματεύσει ω παρατηρητή. Όχι ε, μόνο μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, αλλά και σε κάθε περίπτωση όπου θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις για ε, την ευρωπαϊκή ε, αγορά ενέργειας και για την ε, διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, τη συνάδελφο για τις παρατηρήσεις, ο κύριος Σιλικιώτης, εκ μέρου της ΕΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γκραντζοντεύσκη για την εισήγησή του. Παρόλο που πρέπει να πω από την αρχή ότι ω ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά έχουμε διαφορετική θέση για το πώς πρέπει να διαμορφώνονται οι διακυβερνητικές συμφωνίες. Για μας είναι ξεκάθαρο πώς απαιτείται ενισχυμένο κρατικός έλεγχος και εθνική ευελιξία. Δεν γίνεται τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να υπογράφουν διακυβερνητικές συμφωνίες χωρίς την έγκριση της Κομισιός, όπως ζητείται στην πρόταση που έχει καταδεθεί. Ούτε είναι παραγωγικό να είναι υποχρεωτική ακόμα και εκ των προτέρων αξιολόγηση των συμφωνιών από την Κομισιό. Το δε χρονικό περιθώριο που προτείνεται να έχει στη διάθεση της η Κομισιό μέχρι να αποφασίσει για την σοβαρότητα των διακρατικών συμφωνιών είναι υπερβολικά μεγάλο και μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τη συμφωνία που πέτυχαν τα κράτη. Το έχω τονίσει πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην ενεργειακή τροφοδοσία ενώ πολλά κράτη και περιοχές της Ένωσης είναι ακόμα απομονωμένες από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ επικίνδυνο να προωθούνται πολιτικές που περιερίζουν τα, κρατικά, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, αλλά και τη δυνατότητά τους να διαμορφώνουν πολυδιάστατες και αποδοτικές διακυβερνητικές ενεργειακές σχέσεις. Οι προτάσεις που ζητούν αύξηση των εξηγιών της Κομισιόν και μεγαλύτερη εμπλοκή τη στη διαδικασία ακόμα και πριν τη σύναψη των διακυβερνητικών συμφωνιών, είναι προβληματικέ και εμπερικλείουν μεγάλου κινδύνου. Εξίσου προβληματική είναι και η πρόταση τα κράτη-μέλη να είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Κομισιόν ακόμα και για την πρόθεσή του να αρχίσουν διαπραγματεύσει, καθώ και η πρόταση τα αιτήματα των κρατών μελών για εμπιστευτικότητα όσον αφορά σημαντικέ προφορίες να μην περιορίζουν την πρόσβαση τη Κομισιόν σε αυτά. Ιδιαίτερα απαράδεκτη όμω θεωρούμε την προσπάθεια χειραγώγησης των κρατών μελών από την Κομισιόν με την πρόταση που προωθείται για έλεγχο ακόμη και των μη δεσμευτικών πράξεων όπω είναι τα μνημόνια συνεργασία, οι υπουργικέ κοινέ δηλώσει και κοινέ δράσει αναφορικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό ή την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Δυστυχώ όλε αυτέ οι προτάσει μετατρέπουν τα κράτη-μέλη σε πιόνια πλήρω εξαρτημένα από την Κομισιόν καθώς κάθε ενέργειά τους θα προποθέτει πλέον τη σύμφωνο γνώμη της. Αυτό για μα είναι ανεπίπλεπτο. Αντί αυτού τονίζουμε πως θα ήταν ωφέλιμο η Κομισιό να, να έχει ενισχυμένο συμβουλευτικό ρόλο εφόσον όμως ζητηθεί βοήθεια από τα κράτη-μέλη. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι τροποτελεγγύες που καταθέσαμε και ευελπιστούμε πως θα συμπεριληφθούν κάποιες από αυτές τις συμβατικές προτάσεις ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Ο Σάφος Μπορέλη από την πλευρά του EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέω εξ αρχής ε, ότι η δημιουργία μιας ε, πραγματικής ε, κοινή ενεργειακής πολιτικής που θα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της ενέργειας θα ήταν κάτι πολύ θετικό για τους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για να υπογραμμίσω τους λόγους και τις αρχές που διέπουν τις τροπολογίες μας. Εμείς θελήσαμε μέσω των τροπολογιών να αποσαφηνίσουμε το ρόλο της Κομισιόν, αποσαφηνίζοντάς τον, διότι στο αρχικό κείμενο, κατά την άποψή μας, ε, παραμένουν πολλά θεά σημεία. Θελήσαμε να καθορίσουμε ε, σε ρόλο συμβουλευτικό τον ρόλο της ε, Κομισιόν, έτσι ώστε να μην γίνει τρίτος παράγοντας διαπραγμάτευσης, γιατί θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι αυστηρά προκαθορισμένος ο ρόλος των εμπλεκομένων. Εδώ δεν είναι σαφές το κείμενο Επίση, Επίσης, ε, για να αποσαφηνίσουμε το σημείο αυτό, θελήσαμε να ε, υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει η στήριξη της Κομισιόν να είναι καθαρά νομικής φύσεως. Επίσης, ε, θελήσαμε να υπογραμμίσουμε ότι κύριοι πρωταγωνιστές θα είναι οι εμπλεκόμενοι από πλευρά κρατών και στο ρόλο του αυτό θελήσαμε να τους υποστηρίξουμε. Ο επιχειρησιακός, η επιχειρησιακή συμβολή της Κομισιόν θα πρέπει να αφορά και την ενίσχυση του ρόλου των κρατών Σημειώνουμε ότι ε, θα πρέπει η Κομισιόν ε, να έχει συγκεκριμένο ρόλο ε, για συγκεκριμένα όμως θέματα και όχι ε, να αφήνει φες ζώνες όπως γίνεται στην, ε, Κομισιόν, στην ε, πρόταση της Επιτροπής. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το, τα θέματα της προμήθειας ας πούμε δεν, που είναι πολύ πιο μικρό από το στοιχείο που αφορά τις διάφορες χώρες μέλη. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει όταν μια συμφωνία κρίνεται σωστή από όλες τις πλευρές ε, και εάν δεν αντιτίθεται στην ε, ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προχωρά και σαν έλεγχο της συμβατότητας μονάχα και της συμμόρφωσης θα, μπορούμε, θα μπορούσαμε να δεχθούμε το ρόλο της Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει όμως ο ρόλος της δεν μπορεί να είναι εναλλακτικό του ρόλου των κρατών μελών ούτε θα πρέπει να έχει μια τέτοια πρόθεση. Θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσουμε τις αρχές αυτές γιατί διαφορετικά θα έχουν την αίσθηση όλο και περισσότεροι οι πολίτες μας ότι μία μακρινή ε, ε, ε, ανεξέλεγκτη γραφειοκρατία είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σοπχάουζερ, ε, ΙΕΝΕΦ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας, τα κράτη έχουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα για τις διακυβερνητικές ε, συμφωνίες ε, θα πρέπει να έχουν την κύρια αρμοδιότητα ε, διότι πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες χρήζουν της στήριξης των κρατών. Η αρχή της επικουρικότητας αλλά και αυτή της αναλογικότητας μας υποχρεώνουν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα λόγο, ρόλο δεν μπορεί να παίξει σε αυτές τις συμφωνίες που αφορούν την ενέργεια. Η διακυβερνητική διάσταση είναι αρκετή και η Βεβαίως έχουμε και την ενεργειακή ασφάλεια η οποία βασίζεται ε, στα κράτη. Ε, πρόκειται για μια μακρόχρονη ε, πολιτική η οποία αφορά την αποδοτικότητα και την προμήθεια. Εάν προσθεθεί στα κράτη-μέλη η Κομισιόν, προστίθεται στην ουσία η αστάθεια την οποία έχουμε γνωρίσει μετά από την παρέμβασή της. Η ενεργειακή αλυσίδα βασίζεται στις διακυβερνητικές σχέσεις και την επικουρικότητα δυστυχώς οι προτάσεις του συναδέλφου και φίλου ε, εισηγητού επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη θέση της Κομισιόν. Η δυνατότητα εξακρίβωσης εξάντε εκ των προτέρων των συμφωνιών ε, και η ε, μετάδοση των μη δεσμευτικών εργαλείων αφορά, αφορά ανάμειξη της Κομισιόν στα εσωτερικά των κρατών. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι το, τα κοινοβούλια της Μάλτας, της Γαλλίας, Τη ε, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας ήδη ε, καταδικάζουν το κείμενο αυτό ε, λέγοντας ότι καταπατά την επικουρικότητα. Επίσης, τα ποσοστά ε, είναι πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή δεν αφορούν το 34% αλλά 13%. Εάν δεν αφαιρέσουμε το South Stream πέφτουν στο 8% και επομένως είναι δυσανάλογη η προσπάθεια της Κομισιόν και οπωσδήποτε ανώφελη, ε, ε, άχρηστη και οπωσδήποτε αντίθετη με την αρχή της διασφάλισης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, στρέφομαι τώρα στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, Hans von Stell, επικεφαλή τη μονάδα τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, καλή έκθεση και να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έκαναν χρήσιμα σχόλια και υπέβαλαν ε, καλές τροπολογίες. Από την πλευρά της Κομισιόν θεωρούμε ότι, ε, ε ότι η θέση του Κοινοβουλίου καθίσταται αρκετά σαφής ε, και καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θέλει και οδηγείται προς μια φιλόδοξη προσέγγιση βάσει και της πρότασης της Κομισιόν. Δεν θα μπω σε πολλέ λεπτομέρειες όσον αφορά τι διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ίσως όμως ε, θα έπρεπε να υπενθυμίσω τον λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται τώρα να αναθεωρήσει την ε, νομοθεσία σύντομα μετά την αρχική της έγκριση και υιοθεσία. Ε, διαπίστωσε η Κομισιόν ε, ότι δεν λειτουργεί ε, το θέμα αυτό, κυρίως όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες. Ένα τρίτο των διακυβερνητικών συμφωνιών δεν παρέχει την απαραίτητη συμμόρφωση. Το ίδιο συμβαίνει δε και με ένα μεγάλο τμήμα των μη δεσμευτικών πράξεων. Όσον αφορά την εξάντεκ των προτέρων αξιολόγηση, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων. αυτό που θεωρούμε εμείς πολύ σημαντικό είναι να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία, πράγμα που σημαίνει ε, τα, από τη μία το, το δικαίωμα που έχουν τα κράτη-μέλη να συνάπτουν διακυβερνητικές συμφωνίες, γιατί βεβαίως αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες τελικά συμμορφούνται ε, με την ενωσιακή νομοθεσία. Όπως έχει καταδειχθεί ήδη υπάρχουν πολλές ε, λεπτομέρειες οι οποίες μαζί με την διαδικασία διαδικασία ε, εξάντε ε, ε, αξιολόγησης ε, που λέω θα μας οδηγήσουν στο να αξιολογήσουμε τις μη δεσμευτικέ πράξεις και να δούμε ποιος θα είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να αναμειχθεί η Κομισιόν στο σημείο αυτό. Επίσης θα ήταν πολύ ικανοποιητικό εάν μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα οι τριμερείς διάλογοι, πράγμα που θα μας επέτρεπε να δούμε ε, αυτήν την νομοθεσία σαν ένα από τα ε, πρώτα και πολύ σημαντικά παραδοτέα όσον αφορά το γενικότερο θέμα της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Βεβαίως, εμείς θα θέλαμε να διατηρηθεί η φιλόδοξη προσέγγιση και φυσικά να παίξει ο καθένας επικοδομητικό ρόλο στους τριμερείς διαλόγους που θα ξεκινήσουν ως ονούπο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος. Επιστρέφουμε ε, στον ε, εισηγητή μας. Θα ζητήσω λοιπόν από τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Κράσνοντεύσκη, να μας κάνει τις τελευταίες του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν το λόγο. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας οι οποίες ε, επιβεβαιώνουν ε, την ελπίδα μου ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις. Θα ήθελα όμως να σημειώσω και κάτι άλλο. Πρόκειται για ένα ε, θέμα πολιτικής φύσεως. Ε, υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί ε, Στι δηλώσει των συναδέλφων όσον αφορά τι αρμοδιότητες των κρατών μελών, όσον αφορά ε, την ε, ανεξαρτησία των κρατών μελών. Υπάρχουν φόβοι που εκφράστηκαν, δηλαδή φοβούμαστε μήπως παραχωρήσουμε υπερβολικά πολλά τα κράτη-μέλη, μήπως δώσουν πολλές αρμοδιότητες και παραχωρήσουν υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ εκπροσωπώ μια πολιτική ομάδα η οποία ε, αποδίδει μεγάλη σημασία εις ε, την ε, εθνική στην εθνική κυριαρχία και αυτό σχετίζεται και με τη θέση μας όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια δηλαδή καθόλου δεν πρέπει να ξεχνάμε την εθνική κυριαρχία μιλώντας για την ενέργεια θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να μην το λησμονούμε βεβαίως δεν μπορούμε πάντα να συμφωνούμε όλοι σε όλα Ε, κυρίως όταν μιλάμε για την ε, ασφάλεια ε, διαφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης όταν μιλάμε για την αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να δυναμητίζεται η αλληλεγγύη μας όταν μιλάμε για θέματα διασφάλισης της ενεργειακής ε, απόδοσης ε, γιατί ε, θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξουν μπορούν να υπάρξουν κάποια ε, ασθενή σημεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέσω των διακρατικών ε, συμφωνιών και των άλλων πράξεων να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με την, ενεργειακή ασφάλεια. Πρόεδρος, ναι βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι, μια συζήτηση κομβικής σημασίας όπως και εσείς το αναφέρατε. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι στην Επιτροπή η Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 13η Οκτωβρίου, ε, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για το, τους κανόνες που διέπουν τις αγορές περιαγωγής χονδρικής. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, ξέρουμε ότι από τον επόμενο Ιούνιο θα έχουμε ε, μια νέα κατάσταση όσον αφορά την ε, περιαγωγή. Να μην λησμονούμε επίσης ότι έχει ότι έχουμε και την, τον κανονισμό της 15ης Ιουνίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις αγορές περιαγωγής χονδρικής από πλευράς της Κομισιόν Επίσης ε, έχουμε και την, ε, τον οργανισμό TSM, ο οποίος αναφέρει ότι ε, από την 15η Ιουνίου του 2017 δεν θα υπάρξουν πλέον, θα, θα καταργηθούν οι επιπλέον χρεώσεις σχετικά με την περιαγωγή. Από τον ε, Ιούνιο λοιπόν του 2015 θα σταματήσουν οι επιπλέον ε, χρεώσεις χονδρικής ε, περιαγωγής. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε τους κανόνες που διέπουν τι τις αγορές περιαγωγής χονδρικής. Η κυρία Κουπούλα Νάτρι ήδη τον, μάλλον θα, θα συζητήσει την έκθεσή της μαζί μας την 12η Οκτωβρίου, τώρα χωρίς κείμενο θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, η γνωμοδότησή μας, έτσι ώστε να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις σε σχέση με ε, την περιεγωγή χονδρικής. Θα δώσω το λόγο στην αγαπητή Πέτρα Κομπούλα Μάτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ ήρθατε. Νομίζω ότι είναι καλή χρονική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει ότι μπορεί να ε, είναι ταχύτατο και να τηρήσει τι υποσχέσει προ του καταναλωτέ ότι μέχρι την επό... το επόμενο καλοκαίρι δεν θα υπάρχει περιαγωγή, δεν υπάρχουν τέλη περιαγωγή ε, και πρέπει να υπάρξουν βέβαια κανόνε προκειμένου να είναι έτοιμη η περιαγωγή χονδρική ε, Θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ότι καλό είναι να εκφράσουν σήμερα την άποψή τους, ε, όμως πρέπει να περιμένουμε την ε, έκθεση Μπέρεκ ε, και θα ήθελα να, να δω τη δική του απόφαση πριν πάρουμε εμείς τη δική μας απόφαση, γιατί είναι πολύ συνδεδεμένα αυτά τα πράγματα και έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον, στις αγορές. 90 ημέρες ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Αρχίσαμε Καταρχά ε, για τα μηνύματα κειμένου όταν ε, το TSM ε, αρχίσαμε να το συζητούμε. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Πρέπει να υπάρξει, να έχουμε την απόφαση μπροστά μας πριν αρχίσει ο τριμερής διάλογος. Η ψηφιακή αγορά είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ, πρέπει να ολοκληρωθεί, χρειαζόμαστε τι επενδύσει, χρειαζόμαστε τι θέσει απασχόληση και μια ψηφιοποιημένη Ευρώπη. Συνεπώ αυτό είναι ένα μικρό νομοθέτημα το οποίο ε, οδηγεί προ αυτή την κατεύθυνση και όπω είπε και ο πρόεδρο, έχουμε αποφασίσει ήδη, έχουμε ήδη ε, υποσχεθεί στον καταναλωτή ότι θα προχωρήσουμε ε, χρειάζεται μία αναθεώρηση της περιαγωγής χοντρικής και ε, αυτό πρέπει πράγματι να γίνει. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφής. Τρία, τρία ε, όρια τιμολόγησης. Ε, τρία πράγματα. Είναι αυτό επαρκές? Ε, μάλλον όχι, γιατί θα υπάρξει lobbying προς όλους σας από διάφορους φορείς και θα ήθελα να έχω ολόκληρη την ευρωπαϊκή εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να έχουν τα πράγματα. Ευχαρίστω να εξετάσουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την ε, μελέτη αξιολόγησης που καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη έχει γίνει με μεγάλη προσοχή. Βέβαια αμφισβητείται από κάποιους, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου ε, μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί ως βάση, ως αφετηρία. Τα τρία νούμερα μπορεί να είναι πολύ ψηλά για κάποιον, πολύ χαμηλά για κάποιον άλλον. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να ε, υπάρξει ένα συμβιβασμό. Όμω από πολιτική απόψεω ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μα τον καταναλωτή. Υπάρχει το θέμα τη χρήση δεδομένων στο πλαίσιο μια ανταγωνιστική αγορά. Νομίζω ότι η τιμή των δεδομένων είναι το πιο σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ότι η χρήση δεδομένων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αν προσπαθήσουμε να πούμε ότι δεν θα αυξηθεί ή ότι δεν θα έπρεπε, τότε καταστρέφουμε τον ευρωπαϊκό ε, πλούτο και το μέλλον, ε, γιατί πρέπει να υπάρξει η ψηφιοποίηση της Ευρώπης. Όσον αφορά την υπόσχεσή μας προς τον καταναλωτή, αν η τιμή δεν είναι η σωστή, θα θεωρηθεί ενδεχομένως ότι οι καταναλωτές ε, θα θεωρήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεχωριστά μέτρα και σταθμά για τους ταξιδιώτες. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσους ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και εμείς ε, ταξιδεύουμε πάρα πολύ. Πάνω από 90 ημέρες ε, μένουμε στην, στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα. Αλλά για μένα η χρήση των δεδομένων ε, διασυνοριακά σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να μπορεί να στέλνει τα email του και να παραμένει συνδεδεμένος. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα, είναι σαν να του ζητά κάποιος να σταματήσει τη δουλειά του. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια καλή τιμή και απαλλαγή από την περιαγωγή και πρέπει και ο τομέας της χονδρικής να δει σε ποιο επίπεδο ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ε, η τιμή. Έχει, έχει μειωθεί και τα καλά νέα είναι ότι θα συνεχίσει να μειώνεται γιατί δεν είναι γραμμική η κατάσταση. Όσο γίνεται μεγαλύτερη επένδυση και υπάρχει μεγαλύτερη χρήση δεδομένων, δεν είναι πια ίδια η τιμή αναμονάδα. Περισσότερη επένδυση σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι χρήστε και αν είναι περισσότεροι χρήστε μπορεί να είναι φθηνότερη η τιμή αναχρήστη. Αυτό έχει συμβεί ω τώρα και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να επενδύσουμε σε όλη την Ευρώπη στα δεδομένα. Είναι μόνο ένα συγκεκριμένο, μόνο ένα τμήμα τη περιαγωγή, είναι όμω το πιο σημαντικό δεύτερο τμήμα μάλλον, γιατί πρώτα είναι η υπόσχεση προς τους καταναλωτές ε, και να είναι απλούστερη η κατάσταση για τους καταναλωτές και μετά έρχεται αυτό που μόλις είπα. Η εμπιστοσύνη επίσης πρέπει να ε, εξακολουθήσει να ευίσταται. Υπήρξε πολύ, ε, πολλή νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει αυτή η τιμολόγηση να μην έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο κάποιων ε, παικτών από την αγορά, γι αυτό, γιατί αυτό σημαίνει λιγότερος ανταγωνισμός, ε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έξυπνοι καινοτόμοι και νέοι παίκτες ε, να εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά, ώστε να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο ανταγωνιστικότητας αν ε, η περίοδος των 90 ημερών δεν ε, είναι επιτυχής ε, και αν η τιμολόγηση θα είναι σωστή. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την μόνιμη περιαγωγή. Πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας κατά της κατάχρησης ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία και αυτό πρέπει να, το, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παραμένει ισορροπημένο. Πρέπει να πω ότι ε, είναι γεγονός ότι δεν θα έπρεπε η επικοινωνία να σταματά, όπως ακριβώς δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να σταματούν στα σύνορα. Ε, αυτό είναι μια πολύ καλή παρουσία, ε, παρομοίωση. Συγγνώμη, υπερεύει το χρόνο μου κατά ένα λεπτό σχεδόν ήδη. Ναι, λέει ο Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα εισαγωγικά σας σχόλια όσον αφορά την σημασία των κανόνων των αγορών ε, περιαγωγής χονδρικής ε, εκ μέρους ε, του ΕΛΚ, ο σκιώτης της κ. Ρούμπιχ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα γιατί βέβαια περνάμε από την ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών σε μια ενιαία ψηφιακή πλέον αγορά. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί θα πρέπει από τη μία πλευρά να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών ε, και από την άλλη ε, να ε, επιτρέψουμε τις ταχείες επενδύσεις εδώ και την ταχεία εξάπλωση των σχετικών υποδομών. Μέσω της πολιτικής που έχουμε εφαρμόσει έχει δημιουργηθεί πολύ ψηλός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ε, σε αυτόν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και βέβαια αυτό μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένας τέτοιος υγιής ανταγωνισμός. Κατά συνέπεια λοιπόν η δημιουργία αυτής της νέας ευσυχιακής αγοράς αποτελεί την προτεραιότητά μας και από εκεί και μετά οι ε, μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα μπορούν να απορροφήσουν το σχετικό ε, κόστος. Υπήρξαν ε, ε, υπήρξαν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ε, μπόρεσαν να εξαπλώνουν σε όλο του ε, το δίκτυο το σχετικό κόστος χωρίς να υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος. Αλλά το ζητούμενο βέβαια εδώ είναι οι νέες επιχειρήσεις που έχουν εισέλθει στον τομέα και οι οποίες ακριβώς έχουν διασφαλίσει την ύπαρξη ενός υγιούς ανταγωνισμού σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι και στο μέλλον θα είναι θεμητός αυτό ο ανταγωνισμός και είχα αναφέρει και στο παρελθόν ότι εδώ η χοντρική, το κοντριμπόρου σε αυτό το τομέα λαμβάνει η χώρα και μέσω τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ είχα κάνει την ε, σχετική πρόταση η οποία δεν ε, εφαρμόστηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσουμε τώρα είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για αλλά να περάσουμε πλέον στην διαπραγμάτευση τιμών σε ό,τι αφορά ευρώ ανά gigabyte. Γιατί βέβαια ε, κάτι τέτοιο είναι, συμβαδίζει και περισσότερο με τα όσα συμβαίνουν τη σήμερα ημέρα, αλλά και προβλέπει τα όσα, τις εξελίξεις αν θέλετε στο μέλλον. Δηλαδή και ε, στις ίδιες τις χώρες στι ε, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι διάφορες αυτές επιχειρήσεις ε, αναφέρουν τις τιμές τους σε ευρώ ανά γιγαμπάιτ και όχι μεγαμπάιτ οπότε αυτό θα πρέπει να ισχύει και στις τιμές περιαγωγής. Τώρα υπάρχουν βέβαια και διαφορές μεταξύ των net receivers όπως λέγονται και των net senders. Ε, τώρα, ε, για τις ήδη ε, εδρεωμένες επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα, αλλά για τους νέους παίκτες στην αγορά αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα και θα πρέπει να διασφαλίσουμε από την πλευρά μας ότι υπάρχουν ίσοι κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή μεταξύ των ήδη εδρεωμένων επιχειρήσεων και των νέων παικτών, έτσι ώστε ο ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εδώ θα παραμείνει υγιή και θεμετός. Εκείνο που βέβαια είναι το ζητούμενο είναι ε, τα σχετικές, οι σχετικές αυτές υπηρεσίες ε, που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Χέγκερ έχει τώρα το λόγο που τον κύριο Τωσανόφσκι εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Τζουνόφσκι δεν μπορεί να είναι εδώ, ε, δυστυχώς, ε, γιατί άλλες, έχει άλλε πολιτικές υποχρεώσει. υποχρεώσεις. Ε, μου ζήτησε να σα υπενθυμίσω ότι η εισαγωγή της αρχής περιαγωγή χωρίς τέλος την επόμενη χρονιά θα είναι το επιστέγασμα μιας επιτυχούς προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή των τιμών των αγορών χωρών ε, ε, περιεγωγής ε, χοντρικής συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία ταχύτατα με το, Ευρωπαϊκό, με το Συμβούλιο και ότι πρέπει να μειωθούν αυτά, αυτές οι τιμές. Είναι πεπισμένο ότι ο νέο κανονισμό πρέπει να σέβεται την κατάσταση στα κράτη-μέλη και πρέπει να βασίζεται σε απαληθευμένα δεδομένα για το απαραίτητο κόστο των φιλοξενούντων ε, φορέων. Δεν πρέπει να είναι εις βάρος ε, του ε, φορέα που θα επιδοτεί τους φιλοξενούμενους στο δίκτυο. Ανησυχεί λοιπόν για τα μηνύματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτω του κόστους υπηρεσίες δεδομένων για κάποιους φορείς και γι' αυτό θα ήθελε να επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα. Επίσης, ε, αναμένει επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, από τους ε, φιλελεύθερους, ο κύριος Πέτερσεν, που αντικαθιστά τον κύριο Ρόντε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις εκ μέρους του ε, συναδέλφου. Η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ ε, σημαντική θα είναι μεγάλη πρόκληση και ελπίζουμε να υπάρχει καλή συνεργασία με τον εισηγητή που θα οδηγήσει σε ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή της απαγόρευσης των τελών περιαγωγής από τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Όμως αυτή η πρόταση θα πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική με ε, την πολιτική ε, αποτυχιών ε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προθεσμία το, του Ιουνίου 2017 θα γίνει σεβαστή. Ελπίζουμε να υπάρξει μια, ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ του δίκαιου ανταγωνισμού των αναγκών των φορέων και των καταναλωτών και ε, σε αυτό το πλαίσιο αναμένουμε συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπορέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εξ ονόματος Εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ε, σωστή, ε, ε, μια σωστή αγορά κινητής τηλεφωνίας χωρίς διαφορετικές χρεώσεις περιαγωγής, πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είναι η Κομισιόν πιο φιλόδοξη. Η παρούσα πρόταση της Κομισιόν ε, για την μείωση των επιπλέον χρεώσεων στην περιοχή χονδρικής ε, δεν ε, είναι αρκετή έτσι ώστε να μειώσει σε όλους μεγάλους και μικρούς operators την, τη χρέωση. Θα πρέπει να υπάρξουν προσφορές σε κάθε επίπεδο και χωρίς να περιμένουμε μάλιστα μετά από την εφαρμογή της Συμφωνίας για την περιαγωγή αύξηση των τιμών. Πιστεύουμε ότι σε σχέση με τις ε, ε, υπηρεσίες που παρέχονται σε εθνικό επίπεδο ε, δεν είναι ικανοποιητική κίνηση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δέκα φορές επιπλέον χρεώσεις στην χονδρική και επομένως τα περιθώρια εκτόσεων είναι πάρα πολύ και Είναι πολύ μεγάλα. Στην Ιταλία ας πούμε στην το κόστος ε, της ε, μετάδοσης δεδομένων κοστίζει 31 ε, cents το κατά megabyte. Ε, τη στιγμή λοιπόν ε, που η Κομισιόν λέει ότι η οροφή θα είναι 85 cents, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Το σημαντικό είναι να μην πιεστεί ο καταναλωτής έτσι ώστε να σταματήσει την σύνδεσή του στο δίκτυο του διαδικτύου. Στις 15 Ιουνίου του 2019 2017 είναι γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις ε, στις, ε, στην περιαγωγή, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να μειώσουμε πρώτα τις χρεώσεις χονδρικής. Γι' αυτό λοιπόν εγώ και για την μετάδοση δεδομένων αλλά και για τις κλήσεις φωνής θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ, εξ ονόματος του κυρίου Φοντάνα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, του σχέδιου του συναδέλφου Φοντάνα θα ήθελα να πω δύο λόγια. Η κατάργηση ε, των ε, υπερχρεώσεων της περιαγωγής οπωσδήποτε θα βοηθήσουν να θα, θα συμβάλλουν λέω στην καλύτερη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς, αλλά ε, ο κανονισμός από μόνος του δεν μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής. Δεύτερον, Ο κύριος Φοντάνα λέει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί θα είναι σαφείς έτσι ώστε να αποφευθούν οποιασδήποτε επιπλέον χρεώσεις στους καταναλωτές. Ας πούμε, ε, υπάρχουν operators σε κάποια κράτη-μέλη που ήδη έχουν ε, ξεκινήσει να ζητούν ε, επιπλέον χρεώσεις για επιπλέον, επιπλέον υπηρεσίες. Δεν έχει έννοια να υποσχεθούμε στους καταναλωτές ότι τους παράσχουμε κάποιες δωρεάν ε, ή ε, χαμηλής χρέωσης ε, υπηρεσίες όταν ταυτόχρονα οι operators αρχίζουν να αυξούν, αυξάνουν άλλες παροχές. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να διασφαλίσουμε σωστό και δίκαιο ανταγωνισμό οι περισσότεροι από τους μικρούς operators προβληματίζονται γιατί δεν είναι σίγουροι ότι θα καταφέρουν ε, να επιβιώσουν εάν οι τιμές είναι ε, υπερβολικά χαμηλές. Μην λησμονείτε ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση πολλών μικρών operators. Τέλος, η τωρινή λειτουργία το, της αγοράς περιαγωγής μπορεί ε, να επηρεάσει την ε, ε, γενικότερη εικόνα της αγοράς ε, εάν οι εσωτερικές χρεώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι οι χρεώσεις περιαγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις που κάνετε εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητού. Τώρα θα δώσω το λόγο σε άλλους ομιλητές. Η κυρία Καστίγιο Βέρα. Χάρη στη δικιά σας ε, ε, έκθεση και τις διαπραγματεύσεις για, την, ε, για τους κανόνες, ας πούμε, για, συγγνώμη, λόγω της δικιάς σας έκθεσης για την αγορά τηλεπικοινωνιών έχουμε αυτή την έκθεση για τις επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής. Ναι, όχι, λέει η κυρία Καστίγιο, λόγω της συνολικής εργασίας του Κοινοβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα το πω ισπανικά καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι ελήφθη η απόφαση, αλλά τώρα ε, θα πρέπει να κάνουμε το δυσκολότερο, δηλαδή ε, πραγματικά ε, να σταματήσουν οι χρεώσεις περιαγωγής σε ένα χρόνο, σε μερικούς μήνες μάλιστα θα έλεγα, 15 Ιουνίου του 2017 ε, θα σταματήσουν οι χρεώσεις αυτές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει ε, άμεσα να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το θέμα το οποίο ε, συζητάει η έκθεση αυτή η ε, Κομισιόν ε, έχει, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έχει υποβάλει μια πρόταση. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη. Βεβαίως μπορεί κανείς ε, να δει το θέμα αυτό από τη δικιά του πλευρά, τη σκοπιά της χώρας του, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά παρασάγκας απέχει από το να είναι ε, μια νέα αγορά και αποτελεί το άθροισμα εθνικών ε, αγορών και επομένως ε, η άποψη που έχει κανείς για τη μία ή την άλλη τιμή ή υπολογισμό τιμής είναι κάτι το οποίο δεν θα πάψει να υπάρχει. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η πρόθεση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη. Αυτό είναι το σημείο κίνησης και από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί κανείς να συζητήσει ορισμένα στοιχεία της ε, προτάσεως και των προτινόμενων ε, στοιχείων. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι γενικά είναι ισορροπημένη. Ε, τέλος, πιστεύω ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουμε για τις διάφορες παραμέτρους όταν υπάρχουν ας πούμε, συγκεκριμένες προσφορές κλπ. Ε, σε σχέση και με τη διαπραγμάτευση των τιμών έτσι όπως ε, την προτείνει η Κομισιόν. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χώρος έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την πρόταση και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία των εισηγητή και τους σκιώδης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντελκαστήγιο. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ντίτρικ Γκρούσμαν επικεφαλής ε, της ε, αρμόδιας μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι. Ε, Από την πλευρά της Κομισιόν είναι μεγάλη ικανοποίηση που βλέπει την έκθεση αυτή στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής σας. Αναφέρθηκε ήδη ότι η Κομισιόν ε, και ε, από την στιγμή της ε, πρότασης, της δημοσίευσης της πρότασης κανονισμού έχει ήδη προχωρήσει, έχουν συζητήσει ήδη οι διάφορες ομάδες του Συμβουλίου, τι, τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων ε, της ε, Κομισιόν. Επομένως, ε, είναι σημαντικό που ξεκινάει η συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και ελπίζομαι ότι θα διευκολυνθούν και οι συζητήσεις κατά των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συνομοθετών. Ο κύριος στόχος όλων μας είναι βεβαίως ε, να σταματήσουν ε, οι ε, χρεώσεις. Αυτή είναι η βασική, το βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί και είναι σημαντικό να βρεθούν συμβαστικές λύσεις οι δηλώσει σας ε, ήδη περιγράφουν ε, το κύριο, την κύρια φιλοδοξία ε, και το κύριο διακύβευμα αυτής της εργασίας, δηλαδή ακριβώς την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των, των, του κόστου των ε, των τιμών μάλλον που προτείνουν ε, οι operators, ε, τιμή η οποία θα καλύπτει τις υποχρεώσεις τους και από την άλλη πλευρά να δοθεί δυνατότητα σε όσο γίνεται περισσότερους operators να δώσουν τέτοιου είδους δυνατότητες περιαγωγής για όσο γίνεται περισσότερους πελάτες λιανικής που προέρχονται από την εσωτερική τους αγορά. Θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είναι πεπισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αναλύσεις ε, των ε, στόχων δείχνουν ότι οι στόχοι θα καλυφθούν και ότι τα κόστη καλύπτονται κυρίως όσον αφορά την μετάδοση δεδομένων. Από την άλλη πλευρά έχουν ε, γίνει ε, ε, υπολογισμοί και φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι θα καλυφθεί όχι μονάχα, δεν θα καλυφθούν μονάχα οι ανάγκες των μεγάλων operators αλλά και των μικροτέρων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη βεβαίως την ρήτρα εξαίρεσης για τους ε, μικρούς ε, operators. Τελευταίο σημείο που ήθελα να, πω είναι ότι ε, υπάρχει και η διασύνδεση ανάμεσα τη, ανάμεσα στα προτινόμενα και την επερχόμενη νομοθεσία. Μέχρι το τέλος του χρόνου όλα αυτά τα νομοθετικά στοιχεία θα έχουν καλυφθεί και ε, ε, σύντομα θα δημοσιευθεί και ένα προσχέδιο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε ε, τον Σεπτέμβρη να μπορέσουν όλοι να κάνουν τα σχόλιά τους που ξεκινήσει η διαδικασία επιτροπολογίας. Επίσης, τα παράλληλα έχουμε ζητήσει από τον Μπέρεκ ε, την, ε, μια γνωμοδότηση την οποία θα μας δώσει περί τα μέσα Οκτωβρίου έτσι ώστε τα απαραίτητα στοιχεία, όλα τα απαραίτητα στοιχεία να βρίσκονται ε, στο τραπέζι. Ελπίζω θα τα καταφέρουμε έγκαιρα ε, έτσι ώστε να ε, επιτευχθούν οι στόχοι και οι αρχικές φιλοδοξίες του νομοθέτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητή Μία Πέτρα Κούμπουλα Νάτρη, σας δίνω το λόγο για τις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ ε, όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο και αναφέρθηκαν στα ίδια σημείο ουσιαστικά, πράγμα βέβαια το οποίο ε, σηματοδοτεί μια ε, καλή αφετηρία για την ε, για την περαιτέρω δουλειά που θα κάνουμε εδώ και νομίζω πως ε, και η Επιτροπή αυτό επιθυμεί, δηλαδή να υπάρχει μια καλή βάση για τον τριμερή διάλογο. Που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε την ευρωπαϊκή ε, πτυχή, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή διάσταση όταν εξετάσουμε το τελικό αποτέλεσμα των μέτρων μας. Ε, φυσικά δεν θα είναι καλό ε, να ξεκινήσουμε το φθινόπωρο να συζητάμε τιμολόγια, αλλά επειδή έχουμε υποσχεθεί κάτι στους καταναλωτές μας θα πρέπει να το τηρήσουμε. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι κάτι το οποίο προσφέρει κάποιος εντό τη χώρα του θα πρέπει να είναι σε συγκρίσιμε τιμέ με αυτό που προσφέρει εκτό. Και εδώ ουσιαστικά θα έρθω σε αντίθεση με τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι θεωρούν πως η σημερινή αυτή κατάσταση της διαφοράς δηλαδή είναι θεμητή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους συμπληρωματικές χρεώσεις. Ε, ναι, θα εξετάσουμε λοιπόν, λέει ο το σχέδιο τη έκθεση 12 Οκτωβρίου, η προθεσμία για την υποβολή ε, των τροπολογιών 13 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία εδώ στην Ήτρε θα λάβει χώρα στι 29 Νοεμβρίου. Πάντα σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο, 7 ε, το οποίο μόλι τώρα ολοκληρώσαμε και έτσι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8 τη σημερινή σα διάταξη που αφαίρεται στην χρήση τη ε, ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σας ενημερώσω λοιπόν σε σχέση με αυτό το σημείο ότι ε, συζητήσαμε με την ε, κυρία Πατρίσια Τόια, την πρόεδρο μας ε, και εισηγήτρια αυτής του σχεδίου Εκθεση των λογοζήτημα, τον Ιούλιο και σήμερα θα συζητήσουμε τις 205 τροπολογίες που έχουν υποβάλει διάφοροι συνάδελφοι επί αυτού του σχεδίου έκθεσης όπως γνωρίζετε ε, ο σκοπό εδώ είναι αναθεώρηση μιας, ε, ενός ιδίου πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη ζώνης σηματήτων των 700 MHz. Ε, Μέχρι στιγμή χρησιμοποιείται αυτή η ζώνη για ραδιοτηλεοπτικέ μεταδόσει, αλλά με βάση την πρόταση τη Επιτροπής θα χρησιμοποιείται τώρα για ασύρματε υπηρεσιέ επικοινωνιών. Αλλά βέβαια σε σχέση με όλα αυτά θα ενημερωθούμε από την εισηγητριά μα. Οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Πατρίτσια για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλά κάνατε και αναφερθήκατε στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε για το θέμα αυτό και τις ε, ε, αξιολογήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά το θέμα αυτό. Πρέπει να πω ότι ε, η ανάγκη που ανέφερες εσύ είναι μία ανάγκη την οποία ε, ε, όλοι συμμεριστήκαμε, έστω με διαφορετικές απόψεις, όλοι. Δηλαδή όλοι θεωρούμε ε, ότι η μετάπτωση ας πούμε ε, των ε, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών από, τη, το φάσμα των 700 MHz σε χαμηλότερο δίνει δυνατότητα απελευθέρωσης φάσματος του ραδιοφάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους, πράγμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερος την δική μας Επιτροπή. Γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η οικονομία οικονομία, η παραγωγικότητα στην ε, Ευρώπη ακριβώς ε, διότι θα δοθεί στη διάθεσή της ε, μεγαλύτερο τμήμα του διοδιοφάσματος και επομένως οι καινούργιες δυνατότητες για τους πολίτες κλπ. Επομένως, επομένως ε, η απόφαση αυτή ε, η οποία, της οποίας προηγήθηκε μελέτη ε, και η οποία συζητιέται ακροθυγώς εδώ και καιρό πραγματικά καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας κλπ. Ε, κάναμε την πρώτη συζήτηση, έχουν υποβληθεί 200 τροπολογίες, τις οποίες μπορούμε να ομαδοποιήσουμε ε, πλην ε, μικρών στοιχείων και λεπτομεριών. Οι κύριες τροπολογίες μπορούν να συνδεθούν με 5-6 άρθρα αυτής της απόφασης. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα είναι αυτό που αφορά τη δεσμευτική τροπολογία ε, ε, σχετικά δηλαδή με την απελευθέρωση ε, του φάσματος που θα πρέπει να απελευθερωθεί έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τις επικοινωνίες. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο 2020. Έχουν ε, υπάρξει ε, κάποιες εκθέσεις όπως αυτή η έκθεση Λαμή που αναφέρονται στο 2022. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι θέλουν ε, να βάλουμε ημερομηνία πριν από το 2020 και μερικοί άλλοι οι οποίοι θέλουν ημερομηνία μετά το 2022. η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί ε, μία παράταση δύο ετών, δηλαδή να φτάσουμε στο 2022. Και αυτή ε, ε, θα είναι και μια πρόταση η οποία με βρίσκει σύμφωνη και στη δική μας ε, Επιτροπή, ε, αποδεχόμενη βεβαίως ότι πρώτα απ' όλα ε, θα υπάρξει ένας καθαρός οδικός χάρτης όπου θα, αναφέρεται, θα αναφέρονται καθαρά και οι δεσμεύσεις που θα πρέπει να καλύψουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή δεν είναι μία παροχή χωρίς αντάλλαγμα, αλλά θα είναι μία αντιπαροχή με συγκεκριμένα στοιχεία θα το δούμε και αργότερα και σε σχέση και με ένα άλλο άρθρο, ε, είναι τροπολογίες ε, που ε, ε, προτείνουν ε, συγκεκριμένα δικαιολογητικά και αιτιολόγηση όσον αφορά την αποδοχή της μετάθεσης της ημερομηνίας. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι για αυτά τα δύο επιπλέον χρόνια μπορούμε να αναφερθούμε σε χώρες οι οποίες ας πούμε δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλη αυτή τη μετάπτωση μέχρι το 2020 αλλά υπάρχουν ε, και κάποιες ε, ε, ε, χώρες οι οποίες έχουν πολλές περιφερειακές τηλεοράσεις γιατί δεν έχουμε μονάχα τις, με, τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, τις, τους μεγάλους σταθμούς. Υπάρχουν πάρα πολλές περιφερειακές τηλεοράσεις, περιφερειακοί σταθμοί που θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουν όλοι τα ίδια multiplex, θα πρέπει να αλλάξουν λοιπόν πολλά πράγματα και επομένως χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Άλλωστε είναι δείγμα δημοκρατίας η ύπαρξη μεταξύ πολλών ε, σταθμών, ίσως μερικές φορές μάλιστα είναι και υπερβολικά πολύ και κρίνω από τη δικιά μου χώρα. Μία άλλη ομάδα τροπολογιών αφορά ε, την εμπορευσιμότητα των δικαιωμάτων χρήσης ε, του φάσματος κάτω από τα 700 MHz. Εάν υπάρξει η ε, μετάθεση όσον αφορά ε, την ε, παραχώρηση, την ελευθέρωση, θα πρέπει και να ακολουθήσουν και τα δικαιώματα χρήσης. Τρίτη ομάδα τροπολογιών είναι αυτή που αφορά το εξής. Ορισμένοι συνάδελφοι δεν θέλουν να διαγράψουν το γεγονός ότι Όποιος μπει σε αυτά τα φάσματα θα πρέπει ε, να διασφαλίσει, να εγγυηθεί πρώτα απ' όλα ε, μία ικανοποιητική ε, διάθεση στην εθνική επάρκεια επικράτεια, συγγνώμη. Ε, και επίσης ε, ότι θα ε, δεχτεί τη δέσμευση του άρθρου 3 για 30 ΜΜ. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους operators να διασφαλίσουν αυτήν την ταχύτητα για όλους, γιατί υπάρχουν και τεχνικές δεσμεύσεις. Ε, αυτό λέει η Κομισιόν και πιστεύω ότι και εμείς θα πρέπει σαν Κοινοβούλιο ε, να ε, ζητήσουμε, να ζητήσουμε από τους παρόχους μια καθολική υπηρεσία σε ικανοποιητική ταχύτητα. Θα δούμε από κοντά τις άλλες τροπολογίες και τις λεπτομέρειές τους. Επίσης, για να υπάρχει η διασφάλιση των, ε, ε, ε, των operators ότι θα έχουν σταθερή δυνατότητα χρήσης του ραδιοφάσματος. Ζητούμε τουλάχιστον μέχρι το 2030 να διατίθεται αυτή αυτό το ραδιοφάσμα και αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 5. Πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που ζητούμε τόσες ε, τροπολογίες, τόσες διαφοροποιήσεις μάλλον και τόσες αλλαγές, είναι καλό και είναι δίκαιο να δώσουμε κάποιο αντίβαρο, ας πούμε, κάποια εγγύηση ε, και στους ε, operators, γιατί αυτοί οι οποίοι θα θα επενδύσουν στο φάσμα κάτω των 700 MHz θα πρέπει να έχουν κάποιες ελάχιστες διασφαλίσεις. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο προτείνω ε, να ε, ε, εισάγουμε, αλλά δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι. Ένα άλλο σημείο που δεν βρίσκει σύμφωνο όλους είναι το εξής. Η Κομισιόν λέει ότι κάτω από τα 700 μπορεί να γίνει ένα data link για τους operators. Υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι downlink δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι θα υπάρξει ένα downlink, αλλά με συγκεκριμένα συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις. Μπορούμε να αφήσουμε αυτό το downlink, ε, αλλά ε, εγώ ακόμα δεν έχω διαμορφώσει άποψη. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με τους, με τους σκιώδεις. Επίσης, τι θα γίνει με το φάσμα των 700. Ε, ποιος θα είναι ο δικός ε, χάρτης. Ε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το 2017 θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον οδικό χάρτη ε, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτοποίησεως και ελέγχου των στοιχείων ε, και μετά να δούμε και τις ε, σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, εάν να δούμε δηλαδή το θέμα των παρεμβολών, γιατί γιατί εάν ε, γειτονικές χώρες δεν ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό και δεν σεβαστούν ε, ταυτόχρονες ημερομηνίες ε, θα προκύψει ένα θέμα παρεμβολών. Επίσης, το θέμα της αποζημίωσης των χρηστών ε, που θα πρέπει ενδεχομένως να αγοράσουν ε, διαφορετικούς εξοπλισμούς και κτλ. Εγώ πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό των αποζημιώσεων των χρηστών. Τελευταίο, οπότε θα πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις για την χρήση του φάσματος. Η Κομισιόν λέει 2025, εγώ λέω 2023, έτσι ώστε να προλάβουμε την επόμενη παγκόσμια διάσκεψη. Επομένως, ε, σας είπα ε, γύρω από ποια θέματα ε, περιστρέφονται οι τροπολογίες. Σας είπα και κάποιες δικές μου απόψεις όσον αφορά τις τροπολογίες. Αυτά. 11 λεπτά μιλήσατε. Σε Συγχαρητήρια. Η συγγήτρια μας είπε ότι είναι δυνατόν να υποθεί. Κυρία Ντελκαστή Γιοβέρα, εκ μέρους του κυρίου Χόκμαρκ από το ΕΛΚ. Ναι, εκ μέρους του κυρίου Χόκμαρκ, που είναι ένα, ο σκιώδης εισηγητής μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για τη δουλειά της ε, με το θέμα αυτό ως τώρα. Με χαρά περιμένω τη συνεργασία με την κυρία Τόγια και τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές ώστε να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν και να θέσουμε τα θεμέλια ε, τη, όχι μόνο για, τις κινητές, ε, για την κινητή τηλεφωνία αλλά και για την ε, ψηφιακή ένωση γενικότερα. Απλώς αυτό πρέπει να, να υπάρξει στο σωστό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης ραδιοφάσματος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει, να προσελκύσει επενδυτές στη νέα οικονομία με την ε, γρήγορη ε, επέκταση του ραδιοφάσματος ε, από τα 470 MHz, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει την πιο ανταγωνιστική και πιο καινοτόμο αγορά. Αυτή η πρόταση πρέπει να ειδωθεί υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων. Επομένως, η ευρεία ε, εφαρμογή ε, πρέπει να είναι ε, η λέξη κλειδί κατά τις διαπραγματεύσεις. Να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια εναρμονισμένη εφαρμογή κατά το δυνατόν Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα, ε, για το 2020 θα έπρεπε να παραμείνει ως χρονοδιάγραμμα. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε όμως να μπορούν να καθυστερήσουν ε, ε, δύο χρόνια το πολύ, βάσει ε, πολύ συγκεκριμένων λόγων χωρίς ε, να παρεμποδίζουν ε, τη χρήση του ραδιοφάσματος για, την, για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες για τα άλλα κρατημέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε καθυστέρηση να αιτιολογείται και ότι δεν αποτελεί μέσο για το κράτος μέλος, ώστε να καθυστερεί απλώς την εφαρμογή όσον αφορά τη μίσθωση των δικαιωμάτων ραδιοφάσματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ένα όριο την 30 Ιουνίου του 2022, όμως για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και το ότι θα πρωτοστατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση. Προτείνουμε λοιπόν η, η, προθεσμία για την μίσθωση ε, να οριστεί για το 2021. Όσον αφορά τώρα την κινητή τηλεφωνία και τα MBNOs, ε, η διάθεση των, ε, της ζώνης των 700 MHz θα πρέπει να ενθαρρύνει τον, ανταγωνιστό, τον ανταγωνιστών α, μέσω απαιτήσεων ε, για κοινά δίκτυα ε, και οι εικονικούς ε, φορείς. Οι NBNOs μπορεί να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην ασύρματη επικοινωνία και να εξασφαλίσει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Θα έπρεπε να έχει έναν κύκλο ζωής 30 ετών για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και να δώσει τη δυνατότητα ε, απόδοσης των επενδύσεων όσον αφορά τα έσοδα από την εμπορία των άδειων. Χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου για τους κατόχους αδειών, ε, συγκεκριμένα ε, δικαιώματα ε, που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, γιατί υπήρχε στο TSM μία ε, προϋπόθεση η οποία τελικά αποσύρθηκε γιατί δεν μπορούσαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτήν ε, την πρόταση εκ μέρους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τριμερή διάλογο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν αρκετό χρόνο για να εγκρίνουν και να δημοσιοποιήσουν το εθνικό τους σχέδιο. Η ημερομηνία 36 του 2018 θα πρέπει να αντεπεξέρχεται σε αυτές τις ε, προϋποθέσεις αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθυστερήσει πέρα από το 2020 ο ε, χάρτης πορείας θα έπρεπε να δίνει τη σωστή αιτιολόγηση για την καθυστέρηση και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αποφασίσει κατά πόσο είναι αποδεκτή η αιτιολόγηση αυτή λαμβάνοντας υπόψη ε, την, την άποψη της ομάδας πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πέτερσον, εκ μέρους του κύριου Ρόντε, για δεύτερη φορά. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να τονίσω τρία σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ε, ε, ομάδα των φιλελευθέρων. Καταρχά χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Τα ζητήματα των, του ραδιοφάσματο ε, έχουν τεθεί εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει απόφαση σε διεθνέ επίπεδο να, υπάρχει περισσότερες, να υπάρχουν περισσότερε συχνότητε για την κινητή τηλεφωνία και την ασύρματη επικοινωνία. Η, παρά την ε, επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να το κάνει. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ανασκουμποθούν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπολείπεται των προκλήσεων του 5G ε, και πολλών άλλων ε, τεχνολογικών εξελίσεων. Πρέπει η ε, συνδετικότητα των Ευρωπαίων πολιτών να βελτιωθεί επίσης. Η διάθεση του ραδιοφάσματος πρέπει να εναρμονιστεί. Δεν υπάρχουν σύνορα για τις ε, συχνότητε. Η ψηφιακή αγορά δεν είναι ακόμη πραγματικότητα. Πρέπει να υπάρχει συνοχή, τεχνική εναρμόνιση, να υπάρχουν μέτρα για την ε, συνύπαρξη στο πλαίσιο αυτών των συχνοτήτων, ώστε να ε, ενθαρρύνεται η ε, καινοτομία. Κάτι ακόμη, το χρονοδιάγραμμα που έχει άμεση σχέση, έχουμε χάσει πάρα πολύ καιρό ήδη. Ε, τα κράτη-μέλη είχαν αρκετό χρόνο για να απελευθερώσουν τη ζώνη των 700 MHz και να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις. Το 2020 πρέπει να παραμείνει προθεσμία, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν μιλούμε για ευελιξία, πρέπει να είναι ε, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις απολύτως αιτιολογημένες. Ε, ε, αναμένουμε συνεργασία με την εισηγήτρια και τους ε, υπόλοιπους και τους Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπορέλη από την EFTD. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε από πλευρά της ομάδας μας στην συνεδρίαση των ε, των σκιωδών στα τέλη του μήνα. Ε, για το θέμα αυτό. Είμαι σίγουρος ότι για θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα για όλους δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε ε, συμβιβασμό. Εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογίες για την ε, πλήρη κάλυψη και στις απομακρυσμένες περιοχές της Υπέθρου αλλά και τις νησιωτικές περιοχές. Θεωρούμε ότι μέσω μιας ενδιάμεσης έκθεσης τον Ιούνιο του 2020 2019 θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες ε, ε, ε, ε, ε, καλύτερες, ε, επιδόσεις γιατί δεν είναι δυνατόν εσαΐ να καθυστερούμε την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε οποιαδήποτε καθυστέρηση και επικοδομητικά να συνεργαστούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο γιατί αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη γιατί ξέρουμε ότι το τηλεοπτικό το οποίο σε, ακόμα και στη δικιά μου χώρα ε, είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά θα πρέπει να δούμε, να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα ε, στα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών από τη μία και των απερέτρους από την άλλη. Ε, σε ορισμένες χώρες όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει και, ένα, και την δυνατότητα απελευθέρωσης της, του ραδιοφάσματος και της επιζωνικότητας που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασία και ε, να βοηθήσει την, ε, τον, την ανταγωνιστικότητα στο, στην τροπολογία μας 187 που σχετίζεται με το άρθρο 5 ε, αλλά και με τα άρθρα 2 και 3 αναφέρουμε ε, την διαφάνεια των διαδικασιών. Εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στο θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να, να απαιτήσουμε μεγάλη συνδεσιμότητα για όλους τους πολίτες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με μικρές χαμηλές, ε, ε, χαμηλές τιμές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η χορήγηση ε, αυτής της ζώνης συνοτήτων από τα 470 έως 790 MHz αποτελεί ένα ε, από πολιτικής άποψης ε, λεπτό ζήτημα δικότερα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν δύο πτυχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από τη μία είναι αρμονισμένη προσέγγιση από την πλευρά μας και από την άλλη πλευρά η ταχύτητα της όλης διαδικασίας και αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το χρονικό μας ορίζοντα που έχουμε θέσει δηλαδή ε, για ε, την ε, χορήγηση και την διασφάλιση δικτύου 5G, ούτως ώστε να παραμείνουμε σε ηγετική θέση στον κόσμο. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στην ταχεία εφαρμογή αυτής της αναδιάθεσης της ζώνης συχνοτήτων, εδώ επανέρχομαι στα όσα έχει προτείνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις δεσμευτικές προθεσμίες, ναι, 2000 2020 είναι καταληκτική προθεσμία και 2022 θα είναι η προθεσμία ε, για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θα πρέπει να είναι σαφώς αιτιολογημένο το γιατί έχει χορηγηθεί αυτή η παράταση των δύο ετών. Σε ό,τι αφορά το review, την αναθεώρηση και εγώ ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει αυτή ε, να, να λάβει χώρα πριν από το Παγκόσμιο Φόρτο 2023 και, όχι, και όχι το 2025. μετά, σε ό,τι αφορά τα, την, το χρονοδιάγραμμα που θα δώσουμε στα κράτη-μέλη, ε, Προφανώ για την ε, υποβολή των προτάσεών του θα πρέπει να θέσουμε ε, την κατάλληλη προθεσμία, όπω για παράδειγμα το 2018. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχει συζητηθεί μακρόν αυτό το ζήτημα, οπότε μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο του ρυθμού μα και να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει τελικά και τη σωστή εφαρμογή του roadmap. Δηλαδή να μην φτάσουμε τον Ιούλιο του 2018 να συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο. Τώρα, θεωρώ πως θα πρέπει η, η, η διάρκεια ισχύω των αδειών για την διαχείριση αυτών, για την αξιοποίηση των ε, συχνοτήτων θα πρέπει να είναι στα 30 χρόνια. θεωρώ πως είναι μια πρακτική η οποία ήδη ε, χρησιμοποιείται εκτεταμένα και νομίζω πως θα πρέπει να έχουμε μια ε, λογική προσέγγιση έτσι ώστε δηλαδή να μπορέσουμε αυτή η διαχείριση των αδειών να γίνει με ε, αποτελεσματικό και με ρεαλιστικό τρόπο και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και οι συχνότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Πίλαρ Καστήλο Μαλερ μοίρασε εκ μέρους του κυρίου Χόκμαρκ, ο οποίος με τη σειρά του είχε εκπροσωπήσει άλλους αλλά τώρα εσείς θα λάβετε το λόγο για να εκφράσετε τη δική σας άποψη. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, συνεργαζόμαστε στην ε, Εσκαλώς με αυτούς τους συναδέλφους. Χθες ε, η G20 αποφάσισε να συγκαλέσει συνάντηση των ε, υπουργών ή όσων είναι υπεύθυνοι για την ψηφιακή ανάπτυξη των χωρών ε, του G20, έτσι ώστε να καθοριστούν ε, σχέδια και τρόποι συνεργασίας ε, έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία με τα οποία ασχολήθηκε αυτή η διάσκεψη των G20, δηλαδή πώς να αναπτυχθεί η οικονομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι προφανές ότι ε, η ανάπτυξη της, ε, του φάσματος των 700 MHz ε, και θέματα κάλυψης όπως είναι η μεγάλη ταχύτητα και ε, βεβαίως και η πλήρης ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενεάς είναι κάτι απολύτως επίγον. Σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν, σε σχέση με τη θέση της εισηγητρίας, Πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές βλέπω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, πλην ε, μικρών διαστάσεων απόψεων που πάντα υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα ε, ε, όμως να αναφερθώ σε δύο στοιχεία, ένα που μόλις αναφέρθηκε, δηλαδή η αδειοδότηση των 30χρονη, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, γίνεται πιο ελκυστικό το ζήτημα και επομένως θα, θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κυρίως όμως ε, ε, αναφέρομαι ή στην παράταση από το 20 στο 2020 2022, δηλαδή αυτή η διετής περίοδος ε, για την μετάπτωση ε, του φάσματος. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν, να εγγυηθούν ότι εάν υπάρξει επιμήκυνση σε μία χώρα, μπορούν γειτονικά κράτη να ζητήσουν ε, την ίδια παράταση. αλλά ότι μπορούν ε, να παραμείνουν ε, και σε την ημερομηνία του 2020, γιατί διαφορετικά αν όλοι το ζητούν θα υπάρξει ένα είδος ντόμινο. Εάν επομένως ζητήσει κάποιος την παράταση μέχρι το 22 και του δοθεί, να μην υποχρεωθούν όλοι οι γείτονες ε, ε, να ε, μην σεβαστούν την αρχική ημερομηνία του 2027 και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στην κυρία Κάλλας, την εισηγητρία μας, για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αγορά. Ναι, θα συνεχίσω εδώ τη σκέψη που ξεκίνησε ο συνάδελφος. Δηλαδή, εάν ο στόχος μας εδώ, ε, σε αυτό το φάκελο, είναι να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της ζώνης συνοτήτων των 700 MHz και αφόσον ε, το Συμβούλιο από την πλευρά του έχει συμφωνήσει ότι θα υπάρχει δυνατότητα ε, για ορισμένα κράτη-μέλη να έχουν ε, μια μεταγενέστερη προθεσμία, ε, τότε βρισκόμαστε σε αντίφαση, γιατί δεν υπάρχει ακριβώ αυτή η ενιαία προσέγγιση. Ναι, είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε εξαιρέσει για ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα είναι στη θέση να εφαρμόσουν αυτήν την ε, συμφωνία. Αλλά εάν αυτό ισχύει και θα πρέπει να δέσουμε μια τέτοια ευρύτερη προθεσμία, ίσω θα πρέπει να δώσουμε πιο σύντομη προπραχία προθεσμία για άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εκείνα τα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να επιτύχουν την εφαρμογή το 2020, ίσως θα μπορούσαν να το επιτύχουν και το 2018. Ε, και κάτι ακόμα που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι εάν προβλέψουμε εξαιρέσεις για ορισμένα κράτη-μέλη, δηλαδή μεγαλύτερη προθεσμία, τότε θα πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένου κανόνε που θα διεύουν αυτέ τι εξαιρέσει. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι δεόντω αιτιολογημένη αυτή η παράταση, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα δικαιολογούν μια τέτοια παράταση, όπω για παράδειγμα μη επιληφθέντα ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα ή ε, ζητήματα, ή ανάγκε μετάβαση ε, migration, όπω λέγεται, στι ε, κατάλληλη λογική υποδομή για την λόγω ζώνη συχνοτήτων. Αυτοί οι λόγοι θα πρέπει να αναφέρονται δηλαδή μέσα στον κανονισμό και η Επιτροπή από την πλευρά τη θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή, αν θέλετε, του φορέα διευκόλυνση αυτή τη ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριο Σάνκελ, αντιπρόεδρο. Ναι. Ε, και εγώ ε, έπρεπε να εκπροσωπήσω να μιλήσω εκ μέρου του δικού μα αστυνομικού του Ζαμπασέλ. Οπότε να πω εκ μέρου του ότι από την πλευρά μα από το ECR, εμεί ήμασταν σαφεί ότι μα προβληματίζει σε δύο στοιχεία έχουμε δύο σχόλια να κάνουμε σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή. Χαιρόμαστε για το γεγονό ότι στο σχέδιο τη έκθεση και στι τροπολογίε υπάρχει μια ευρεία συνένεση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά ε, ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, ότι αυτές οι διατάξεις που αφορούν μόνο το downlink για τις συχνότητε κάτω των 700 MHz ε, είναι πράγμα το οποίο εξακολουθεί να μα προβληματίζει. Δεν λαμβάνονται δηλαδή ε, ε, υπόψη οι πρόσφατε εξελίξεις σε αυτό το τομέα, η τεχνολογική πρόοδος και ταυτόχρονα αυτό το μέτρο θα ήταν περιοριστικό και καθόλου χρήσιμο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε ε, κατηγορηματικά κατά των ε, υπηρεσιών downlink. Απλά θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς στον πρόσωπο αυτής της νομοθεσίας. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει ευρεία συνένεση με αυτές τις εξαιρέσεις ε, την παράταση δηλαδή της προθεσμίας των δύο ετών. Ναι, υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την την εφαρμογή και υπάρχει χρησιμότητα για κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμω πλευρά θα πρέπει να σεβαστούμε το γεγονό ότι ε, τα κράτη-μέλη χρειάζονται κάποιο χρόνο για να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την ε, μετάβαση και οι χρήστε ήδη ίδιοι χρειάζονται ε, κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν στι νέε τεχνολογίε. Και αν υπάρχουν δυνατότητε θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία στο κείμενο του κανονισμού για να μπορέσουν ακριβώ να αξιοποιηθούν τέτοιε ευέλικτε δυνατότητε. Πάντω χαιρόμαστε, επιχαίρουμε το γεγονό ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση ό,τι αφορά αυτή την πρόταση του κανονισμού και αναμένουμε με ενδιαφέρον την άλλη συζήτηση που θα κάνουμε με τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε για την εξέβρεση ενό συμβιβασμού. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο του συνάδελφου, την Ακομπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ. Ε, πολύ σύντομα να πω ότι ε, ε, πριν από την ε, συνάντηση ITU θα έχουμε ε, φτάσει στο, στο κείμενό μα ε, σε, ένα συμφωνημένο κείμενο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε λάβει υπόψη μας ε, και άλλες νομοθετήσει σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση των, των 5G. Αυτό μας ανησυχούσε λίγο να μην καθυστερήσουμε πολύ, οπότε πραγματικά είναι καλό το χρονοδιάγραμμα και υποστηρίζω πλήρως το περιεχόμενό της. Την, την περασμένη Παρασκευή στην δική μου χώρα εγώ ήμουν ήδη βέβαια στις Βρυξέλλες, αλλά στη χώρα μου έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των ε, επιχειρήσεων ε, που δραστηριοποιούνται ε, σε αυτό το τομέα, ώστε να διερευνηθεί το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η ζώνη συγχνοτήτων, ειδικότερα προκειμένου το broadcasting, η εκπομπή δηλαδή, οι να μπορούν να αξιοποιηθούν και στο επίπεδο των των κινητών επικοινωνιών. Άρα εκείνο που προσπαθούν να, να επιτύχουν με αυτόν τον τρόπο είναι οι, οι ευρυζωνικές ε, υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω αυτής της ζώνης συχνοτήτων να είναι και κινητές ταυτόχρονα. Αυτό θα πρέπει κάτι τέτοιο να, ε, να, να ισχύει στη σημερινή εποχή, να, να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και αυτή η προσπάθεια και αυτή η πρώτη προσέγγιση έγινε όπως σας είπα την τελευταία Παρασκευή και αυτό είναι καλό. Δηλαδή ότι τελικά αυτή η ζώνη συχνοτήτων δεν είναι περιορισμένη γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά οι διαφορετικέ δηλαδή υπηρεσίε ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ανδρέα Γκάι, ε, ε, επικεφαλή τη ε, μονάδα τη DG Connect τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλησπέρα σε όλου, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου ε, στην εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο ε, της έκθεσης και για όσα ανέφερε ε, προηγουμένως, γιατί πραγματικά υπάρχουν μια σειρά από ισορροπημένα στοιχεία μέσα σε αυτή την θέση. Θα ήθελα εγώ να επιμείνω από την πλευρά μου σε δύο από αυτά, τα οποία ανέφερε και η συγκεκριά. Το ένα από αυτά είναι η διαθεσιμότητα αυτή τη ζώνη συχνοτήτων έω το 2020 και από εκεί και μετά το ζήτημα της ζώνης συχνοτήτων κάτω από τα 700 MHz. Ε, ε, Νομίζω πως είδαμε πω πολλέ ανακοινώσει σε ό,τι αφορά το 5G, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, την τυποποίηση, τα όσα κάνει η Κίνα σε αυτό το τομέα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιαπωνία και ούτω καθεξή, μα δείχνουν ότι είναι σημαντικό αυτή η ζώνη συχνοτήτων να καταστεί διαθέσιμη έως το 2020, αν αυτό είναι δυνατό. Και αυτή η πρόταση που έχει γίνει να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης από την πλευρά τη Επιτροπή για για το 5G, πράγματι για λόγω έκθεση θα δημοσιευθεί από την Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα και θα μπορούμε σούμε, να δούμε εκεί πιο προσεκτικά τι ακριβώ ε, προτείνουμε. Ναι, είναι σημαντικό λοιπόν, εάν θέλουμε να παραμείνουμε εδώ, να έχουμε ηγετικό ρόλο, θα πρέπει η αξιοποίηση να ξεκινήσει μέσα στο 2020. Θα πρέπει να αποφύγουμε καθυστερήσει και κατά τη δική μα άποψη υπάρχουν πολύ περιορισμένε αιτίε οι οποίε δικαιολογούν μια παράταση τη προθεσμία, μια καθυστέρηση για παράδειγμα ε, μια ε, διασυνοριακού χαρακτήρα συμφωνία με τρίτη χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι οποίε ιδιαιτερότητε δεν επιτρέπουν την έγκαιρη εφαρμογή. Υπάρχουν επίση κάποιοι λόγοι θεμητοί για καθυστέρηση. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένα ο οδικό χάρτη θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους. Αναφέρθηκε και η δυνατότητα να προβαίνει σε ένα σχετικό έλεγχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια και οι επιπτώσει τέτοιων καθυστερήσεων, τέτοιων παρατάσεων τη προθεσμία για, για άλλα κράτη-μέλη. Ε, τώρα, εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίε, όπω για παράδειγμα η Ιταλία που αναφέρθηκε, ναι, θα πρέπει να εξετάσουμε. Ε, και να βρούμε λύσεις για αυτά τα κράτη-μέλη. Νομίζω πως υπάρχουν δυνατότητες και στην περίπτωση της Ιταλίας να βελτιώσουμε καλύτερα ε, το, το loading των υφιστάμενων ε, συχνοτήτων, αυτό το multiplexing ε, που ανέφερε μόλις τώρα μια συνάδελφος. Για παράδειγμα, το ζήτημα της προσέγγισης σε σχέση με τους καταναλωτές, ώστε να μην φτάσουμε στο 2020 να έχουμε πολύ υψηλές τιμές για τις σχετικές υπηρεσίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ζώνη συχνοτήτων κάτω από τα 700 MHz και την δυνατότητα ζώνης downlink ή όχι, εμείς συμφωνούμε με τα όσα προτείνει η συγκήτρια, δηλαδή μόνο downlink. Και αυτό γιατί, γιατί ε, μια ισορροπία σε αυτήν την ζώνη συχνοτήτων. Γιατί μας παρέχει και ευελιξία ε, και μας δίνει και μια, μια κατεύθυνση. Και αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να την αποφασίσουμε, να τη χαράξουμε τώρα. Δηλαδή, ε, προκειμένου να μπορέσουμε να, έχουμε την, να επηρεάσουμε την ε, διεθνή τυποποίηση, αλλά και προκειμένου να δούμε προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των 5G. Ε, και ε, η, αυτή η επίδειξη που έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Φιλανδία καταδεικνύει ακριβώς αυτήν την, τις δυνατότητες της τεχνολογίας μόνο downlink. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε τώρα στην εισηγήτριά μας, Πατρίτσια Τόια. Έχετε πάνω από 30 λεπτά. Ωραία, ε! Μα τι λέτε πρόεδρε, εγώ έλεγα να μην μιλήσω καν, γιατί μίλησα πάρα πολύ την πρώτη φορά, στην πρώτη μου παρέμβαση. Εν πάση περιπτώσει όμως, για λόγους ε, αποσαφήνισης ε, και σαφήνειας θα ήθελα να πω δύο λόγια. Θα τα συζητήσουμε ξανά βέβαια τα συμβαστικά, ε, συμβαστικές απολογίες με τους συναδέλφους, των, τους σκιώδες. Εμείς πρέπει να νομοθετήσουμε ε, να νομοθετήσουμε ξέροντας ε, ποιοι είναι οι στόχοι. Στόχος είναι ε, να κινηθούμε γρήγορα έτσι ώστε να δώσουμε ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί, να μην προκληθεί μια αντίδραση κατά της Ευρώπης, δίνοντας την εντύπωση ότι ζημιώνονται οι πολίτες. Όπως έλεγε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, τέτοιου είδους ε, αλλαγές ε, προς την ανταγωνιστικότητα και τα λοιπά μπορεί να προκαλέσουν κάποια, κάποιους προβληματισμούς και αυτούς τους προβληματισμούς θα πρέπει με προσοχή να τους αντιμετωπίσουμε γιατί διαφορετικά ίσως οι πιο ασθενείς πολίτες θα σκεφτούν ότι η Ευρώπη γίνεται όλο και χειρότερη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, και εάν δούμε ότι κάποιος χρειάζεται περισσότερο χρόνο και αν αυτό το αίτημα για περισσότερο χρόνο δεν είναι απλώς δικαιολογία αλλά είναι ανάγκη, θα πρέπει να παράσχουμε το χρόνο αυτό. Όπως πολλοί είπαν, εμείς δεν θέλουμε ε, να δώσουμε αυτήν την δεν θέλουμε να δώσουμε αυτή την παράταση ε, κολλώντας τον τοίχο αυτών που ζητά την παράταση. Ε, αλλά θα πρέπει να δούμε, όπως είπε ο συνάδελφος του ECR, ε, να, να τη δούμε την παράταση αυτή σαν ένα είδος ευελιξίας Το σημαντικό λοιπόν είναι να ξέρει κανείς ότι υπάρχει μια ημερομηνία η οποία είναι προθεσμία στην ουσία και όχι ε, μια ημερομηνία η οποία αυτόματα θα πρέπει ε, να γίνει σεβαστή και ότι εάν ο ένας τη σεβαστεί αυτόματα θα πρέπει να την ε, σεβαστούν και οι άλλοι. Επίσης όταν εγώ λέω ότι μπορούμε να παρατείνουμε μέχρι το 2022 δεν θεωρώ ότι παρέχεται μια εξαίρεση η οποία όμως για να παρασχεθεί θα πρέπει να μελετηθεί με το μεγεθυντικό φακό και σε κάθε λεπτομέρεια. Εγώ την αισθάνομαι σαν μια μεγαλύτερη ευελιξία. Μια ε, ευελιξία λοιπόν η οποία με κανένα τρόπο δεν, ε, δεν κάνει ας πούμε ένοχο ε, αυτόν που ζητά αυτήν την ευελιξία. Εν πάση περιπτώσει όμως με τους συναδέλφους θα ξανασυζητήσουμε το θέμα και θα δούμε λίγο ακόμα και αυτούς που έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση να συνεργαστούμε για να προετοιμάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία λοιπόν στην Ήτρε στις 13 Οκτωβρίου του 2016. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτά. Περνάμε στο επόμενο σημείο της Μερσίας διατάξεως που προβλέπει τα διάφορα. Υπό τα διάφορα δεν υπάρχει κάτι. Ε, σημείο 10 η προσοχή σε συνεδριάσεις. Ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η επόμενη συνεδρίασή μας είναι η 26, την 26 Σεπτεμβρίου 2016 από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ε, ξεκινήσαμε πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και μπράβο μας. Another 10 months in front of us without holidays, almost. Almost. Okay.